Bueno, vamos a empezar, si les parece. Vamos a empezar. Le ruego al staff, por favor. Vamos a empezar nuestra... Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ε, την απογευματινή ακρόαση. Ξέρετε κι εσείς πως πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και που θα μας μιλήσουν ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κεντρική Ασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιφερειακή στρατηγική για την ε, περιοχή και μάλιστα έχει και διμερείς σχέσεις με τις ε, πέντε χώρες που ανήκουν σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Η περιφερειακή στρατηγική αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αναθεώρηση και το Συμβούλιο θα εγκρίνει κάποιες αποφάσεις ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο άμεσο μέλλον. Νομίζω πως η ανταλλαγή απόψεων σήμερα το απόγευμα είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο γιατί γίνονται ερωτήσεις και σε άλλες ε, επιτροπές το θέμα έχει να κάνει με το ποια είναι η πραγματικότητα επιτόπου στην Κεντρική Ασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα βεβαίως είναι μία παράμετρο στην οποία θα πρέπει να αξιολογήσουμε ε, και εμείς μια που είμαστε η αρμόδια υποεπιτροπή. Βεβαίως υπάρχουν ε, όλο και περισσότερα ε, συμφέροντα στην Κεντρική Ασία και είναι μια περιοχή η οποία έχει τεράστια ενεργειακά αποθέματα όπως επίσης γιατί πολλές από τις δικές τους οικονομίες βρίσκονται σε ανάπτυξη, προκλήσεις, θέματα ασφάλειας και όλα αυτά ε, είναι κομμάτι των σχέσεων που έχουμε με την Κεντρική Ασία. Έχουμε έναν ειδικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πίτερ Μπούριαν, ε, που ε, έλαβε τη θέση αυτή στις 15 Απριλίου και ελπίζουμε πως ο δρογερισμός του αποδεικνύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει την περιοχή αυτή του κόσμου στα σοβαρά. Και βεβαίως πώς λαμβάνουμε υπόψη το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεόντως. Έχουμε λοιπόν και τις δικές μας αντιπροσωπείες που ασχολούνται με τα θέματα, αλλά και η δική μας υποεπιτροπή θα παρακολουθήσει στενά το θέμα αυτό. Το πώς λοιπόν εξελίσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε μία από τις χώρες της περιοχής αυτής. Έχουμε κοντά μας άτομα πολύ σημαντικά πολύ ε, ενημερωμένα που γνωρίζουν σε βάθος την κατάσταση της χώρας. Η κυρία Ρίτμαν είναι ε, η πρώτη ομιλήτρια, εκπροσωπεί τη Human Rights Watch και θα μας παρουσιάσει γενικότερα το τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Και μετά θα συστήσω τους ομιλητές έναν έναν ε, για να θυμηθείτε κι εσείς ε, ποιοι είναι και τι κάνουν. Όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να ξεκινήσετε κυρία Ρίτμαν. Λοιπόν, ε, μπορείτε να ακούσετε τα ρώσικα στο 25 για να παρακολουθείτε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Στα σημερινά μου σχόλια θα αναφερθώ στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την προσέγγιση τη κυβερνήσεις Κεντρικής Ασίας για το θέμα αυτό. Όταν υιοθετήθηκε αυτή η στρατηγική το 2007, είχαμε την πρώτη συνολική προσέγγιση για ένα θέμα το οποίο συχνά φαίνεται ξεχασμένο, όπως και η περιοχή αυτή. Ετέθη λοιπόν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προτεραιότητες στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξεκίνησε ένας δομημένος διάλογος με τις κυβερνήσεις της περιοχής για να έχουμε σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Τον Ιούνιο του 2012 οι Υπουργοί Εξωτερικών υιοθέτησαν ένα καινούργιο στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, στο οποίο έλεγαν πως ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου και η δημοκρατία θα ήταν αντικείμενο προώθησης σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης. Ωραία λόγια αυτά, αλλά βεβαίως πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο του τι έχει επιτύχει σε απτό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κεντρική Ασία. Δυστυχώς, όπως υπολογίζει το Human Rights Watch, ούτε η στρατηγική αυτή, ούτε το σχέδιο δράσης ε, έχουν καταλήξει σε μια συνεπή ε, επαφή με τις χώρες αυτές, στις οποίες ε, η κατάσταση είναι προβληματική και επιδεινούμενη. Όπως θα πούν οι λεπτομέρειες, οι συνάδελφοι σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρεια. Η κατάσταση είναι τραγική. Το Τουρκμενιστάν είναι μία από τις πιο καταπιεστικές χώρες. Δεν υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος. Η ελευθερία των ΜΜΕ και της θρησκείας υφίσταται δρακόντιες απαγορεύσεις και υπάρχει ο συνεχής κίνδυνος αντιπίνων από την κυβέρνηση. Η φυλάξη χρησιμοποιείται για πολιτική αντεκδίκηση και για να περιοριστεί το δικαίωμα ταξιδιού του κόσμου στην επέτειο της ε, φαγής του Ατιντζάν στο Ουσμπεκιστάν. Ε, η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχει, υπάρχουν βασανιστήρια όσοι ασκούν τη θρησκεία τους ελεύθερα κοντε εκτός κρατικού ελέγχου και δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης. Τα μέλη της αντιπολίτευσης, οι ακτιβιστές ε, σαπίζουν πίσω από τα κάγκελα με πολιτικές κατηγορίες. Κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάζονται να μαζεύουν βαμβάκι η κατάσταση επιδεινώθηκε στο Καζακστάν μετά τις συγκρούσεις στο Ζανούζεν το 2011. Οι αρχές ε, κατηγόρησαν τους εργαζόμενους στον τομέα του πετρελαίου και ε, φυλάκισαν τον κύριο Καζλόφ ε, της αντιπολίτευσης και έκλεισαν πολλά αντιπολιτευόμενα μήνυε. Το περιθώριο λοιπόν για αντιρρήσεις είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Πέρσι εγκρίθηκαν νόμοι για τα ΜΜΕ και το συνεταιρίζεστε που ε, περιορίζουν την ελευθερία. Η Κυργυζία ξεχωρίζει γιατί το 2010 είχε βουλευτικές εκλογές, όμως εδώ και πέντε χρόνια δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που υπάρχουν στον Νότο, μεταξύ των οποίων ατιμορρησία για τα βασανιστήρια, μετά την βία μεταξύ εθνοτικών ομάδων το 2010. Ο κύριος Ασκάροφ παραμένει επίσης στη φυλακή, φυλακισμένος εισόδια Υπάρχουν επίσης προσπάθειες για να απαγορευτεί η προπαγάνδα των γκέι και να απαγορευτούν οι ξένοι πράκτορες. Επίσης υπάρχουν προβλήματα με τους ΛΟΑΔ. Στο Τατζικιστάν η κατάσταση χειροτερεύει καθώς υπάρχει καταστολή της αντιπολίτευσης. Το 2014 έκλεισαν διάφορα site και απαιτήθηκε η ΜΚΟ να καταγράφουν όλη την ξένη χρηματοδότηση που λαμβάνουν. Υπάρχει συνεχής παρενόχληση και των ΜΜΕ και της ελευθερίας ε, της ε, θρησκευτικής ελευθερίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε ξανά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κεντρική Ασία. Όταν έχουμε τόσο αυταρχικούς ηγέτες δεν φτάνουν τα λόγια. Το πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα για την ε, διαδικασία δημοκρατικής ε, μεταρρύθμισης. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης έχει κρίσιμη σημασία για την κοινωνία των πολιτών. Δημοσιογράφοι και λοιποί εργάζονται με κίνδυνο της ε, ζωής τους για να φέρουν την κυβέρνηση ε, σε θέση να λογοδοτήσει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν απογοητεύονται όταν δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο χρόνο που απομένει τώρα θα ήθελα να αναφέρω τις ανισχύες οργάνωσής μας για την κατάσταση στην Κεντρική Ασία και να τονίσω τους τομεί στους οποίους βλέπουμε πως υπάρχει κάποια ευκαιρία έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί. Παρά τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην ε, πράξη φαίνεται πως τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν περιοριστεί σε κάποιες συζητήσεις μια φορά το χρόνο με τις χώρες αυτές. Οι διάλογοι αυτοί λαμβάνουν χώρα και κλεισμένων των θυρών, χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάζουν τις ε, σχέσεις που υπάρχουν με τις χώρες αυτές. Ε, κατά την άποψή μας υπάρχουν πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημοσιοποιεί συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες έτσι ώστε να είναι σαφής οι προθέσεις της, ε, να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο του διαλόγου και να φροντίσει να παρακολουθείτε η πολιτική σε όλα τα επίπεδα, ειδικά στο υψηλότερο διμερές για να προωθηθούν οι στόχοι που έχουμε. Κανείς δεν αμφισβητεί πως και η ήπια διπλωματία έχει την θέση της. Θα πρέπει να υπάρξει μια πιο ορατή προσπάθεια, ειδικά όταν επισκέπτονται οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της χώρας, για να αναδείξει και την ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σοβαρότητά της. Και έρχομαι άρα στην επόμενη νησία μας. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες προσδοκίες για τις μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέση να αποσπάσει αυτές βελτιώσεις ως μέρος αυτής της διαδικασίας οι διαπραγματεύσει για ενισχυμένε σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν είναι δύο περιπτώσεις οποίε δεν το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σημαντικέ ευκαιρίες. Στην περίπτωση του Καζακστάν η Κάθριν Άστον είχε πει στι ε, αρχές των διαπραγματεύσεων πως θα πρέπει να προωθηθούν οι σχέσει ε, του Καζακστάν. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε δύο ψηφίσματα που ξεκαθάρισαν πω οι ενισχυμένε σχέσει με το Καζακστάν πρέπει να σχετιστούν και να συνδεθούν με βελτιώσει στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και οποιαδήποτε νέα συμφωνία επίση πρέπει να συνδεθεί με πολιτική πρόοδο. Αλλά βεβαίω δεν υπήρξαν τέτοιε μεταρρυθμίσει στο Καζακστάν είχαμε και τον κύριο Καζλόφ και τους εργαζόμενους στον τομέα του πετρελαίου που φυλακίστηκαν, έκλεισαν εφημερίδες της αντιπολίτευσης, ε, κυνηγήθηκαν μειονοτικές θρησκευτικές ομάδες και υιοθετήθηκαν νόμοι που δεν συμφωνούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ποιες μεταρρυθμίσεις ήθελε, οι δηλώσεις πλήν ε, από τις αρχικές της κυρίας Αστών δεν αναφέρθηκαν καθόλου σε αυτά τα θέματα. Τέλος, μια τρίτη ανησυχία ε, είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει τίποτα στην περίπτωση στην οποία δεν υλοποιούνται οι μεταρρυθμίσεις. Για το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να προχωρήσει σε ενίσχυση των σχέσεων αυτών μέχρι να έχουμε πραγματικές βελτιώσεις. Στο πρέπει να υπάρξει σαφέ πρόγραμμα έτσι ώστε η κυβέρνηση να εκπληρώσει τα κριτήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έθεσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών ή αλλιώ να υπάρξουν ρητέ συνέπειε μεταξύ των οποίων και περιορισμοί στη σχέση με την Ένωση. τέλο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει συνέπεια στην στάση τη και να μην επιτρέπει άλλα συμφέροντα όπω αυτά τη ενέργεια και τη ασφάλεια να θέσουν κατά μέρο τη παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν συμβαίνει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει το μήνυμα πως τα πράγματα εξαρτώνται από τις περιστάσεις και αρμιών την αξιοπιστία της. Για το σκοπό αυτό και πριν καταλήξω θα ήθελα να τονίσω τρεις συγκεκριμένους τομείς ανησυχίας που θεωρούμε πως θα μπορούσε να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα η Ένωση. Πρώτον, δεν υπάρχει πλέον χώρος για την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην ελευθερία έκφρασης, ε, του συνεταιρίζεστε και του συνέρχεστε. Πρέπει λοιπόν να επιτραπεί η ειρηνική διαφωνία και να μην υπάρχουν περιορισμοί στην κοινωνία των πολιτών. Δεύτερον, η υπεράσπιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν αυτοί καταλήγουν στη φυλακή με πολιτικές κατηγορίες ε, με βάση άδικες δίκες. Πρέπει να εξασφαλιστεί η απελευθέρωσή τους, όπως, λέγεται και στο, ε, όπως γίνεται στο Ουσμπεκιστάν και στην ε, Κυργιζία. Και το τρίτον είναι να υπάρχει πρόσβαση στις χώρες στις οποίες ε, δεν υπάρχει και να υπάρξει απελευθέρωσή τους η Κυργιζία και η Ουσμπεκιστάν. Θα πρέπει λοιπόν για κάθε μία από τις κεντρές να ακολουθηθεί η στρατηγική τη Κεντρική Ασία και να υπάρχει μια διάφανη διαδικασία για το πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσει με την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι και οι κυβερνήσει αυτέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι υπόλογες απέναντι στην κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. And now, uh, I give the floor. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Γευγένη Ζάφτης, που είναι ένας από τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από τους πιο γνωστούς στο Καζακστάν, δικηγόρος με κύρος, πασίγνωστος για την υπεράσπιση της ελευθερίας έκφρασης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ήδη βρεθεί εδώ στο Κοινοβούλιο με άλλες ευκαιρίες και η σημερινή του παρουσία είναι πολύ επίκαιρη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλύει ακριβώς ε, ε, το θέμα για να προτού συνάψει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με το Καζακστάν. Έτσι θα μπορέσει να μας δώσει τη δική του ε, οπτική που είναι πολύ επίκαιρη σε σχέση με την κατάσταση της χώρας του. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Uh, dear members of the European Parliament, dear guests, <clears throat> thank you for the opportunity to speak here. Which... Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, uh, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε το λόγο σήμερα για να σας μιλήσω για το πρόγραμμα που από κοινού κάνουμε με το Διεθνή Οργανισμό για την Περάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Τουρκμενιστάν ε, και διάφορες άλλες οργανώσεις από το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν. Εγώ θα εστιάσω στο Καζακστάν από όπου προέρχομαι και θα σας δώσω και κάποιες πληροφορίες και για το Καζακστάν και για το Τουρκμενιστάν και για το Τατζικιστάν. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στο Καζακστάν όπω και σε άλλες χώρε τη περιοχή, ε, βασίζεται σε δυναμικές του πολιτικού ε, περιβάλλοντος. Καταρχήν η μετασοβιετική, μετακομμουνιστική ελίτ είναι αυτή που κυβερνά τη χώρα που και βρίσκεται στην εξουσία από το 1989 και κέρδισε τις εκλογές φέτος με πάνω από το 90% των ψήφων με συμμετοχή άνω το 95%. Χαρακτηριστικό αυταρχικό καθεστώς με την ίδια εξουσία εδώ και δεκαετίες. Αυτό το καθεστώς είναι σχετικά ήπιο σε σχέση με το Τουρκμενιστάν και το Ουσβεκιστάν που γειτονεύουν με τη χώρα μας. Αυτό επιτρέπει την ύπαρξη κάποιας πολιτικής αντιπολίτευσης η οποία δεν αντιπροσωπεύεται στο κοινοβούλιο Υπάρχουν κάποια ανεξάρτητα ΜΜΕ, χωρίς ανεξάρτητα όμως ε, ηλεκτρονικά μέσα. Κάποιο χώρο για τις ε, κοινωνίες των πολιτών, ε, για τις οργανώσεις των πολιτών και για κάποιες αντιρρήσεις. Τα ανεξάρτητα ΜΜΕ πρακτικά δεν υπάρχουν και οι επικριτικές, τα επικριτικά site μπλοκάρονται. Η ελίτ αυτή που κυβερνά είναι και η βασική, ε, είναι βασικά εκείνη που, επι, που επωφελήθηκαν από τη μετάβαση από την ε, κρατικο, κρατικοκρατούμενη μάλλον οικονομία στην ε, οικονομία. Ε, της αγοράς. Ε, υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για τον πολιτικό πλουραλισμό, την ισχυρή κοινωνία των πολιτών, ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, δικαιοσύνης κτλ. Γιατί όλες αυτοί οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι απειλή για αυτή την ελίτ. Ως αποτέλεσμα, η κυριαρχούσα ελίτ προτιμά να κρατά τον έλεγχο όλων των κρατικών θεσμών. Δεύτερη παρατήρηση σχετίζεται με την ίδια την κοινωνία. Μετά από δεκαετίες σοβιετικού καθεστώτος και ακόμα και μετά 20 χρόνια της ανεξαρτησίας του Καζακστάν και η κοινωνία του, καθώς και η κοινωνία των υπολείπων ε, κέντροασιατικών ε, ε, κρατών, δεν πιστεύει στην ελευθερία καθόλου. Δεν υπάρχει καμία πρακτική αξία και ο κόσμος δεν θέλει να θυσιαστεί. Για αυτήν ούτε πιστεύουν στις ε, στους θεσμούς βασίζονται αποκλειστικά στο κράτος. Ε, το, τα, τα, τα, τα καθεστώτα αυτά είναι αυταρχικά. Στην περίπτωση του Τουρκμενιστάν είναι μια πραγματική και βίαιη δικτατορία και είναι και ιδιαίτερα διεφθαρμένα όλα τα καθεστώτα αυτά. Ε, να δούμε την κατάσταση του Καζακστάν στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής και θα διαπιστώσουμε ότι είναι λάθος και δεν συμβάλλει, συνάδει με τις διεθνείς αρχές του κράτους δικαίου. Όσο ειδικό, όπως είπε και ο ειδικό απεσταλμένος του ΟΗΕ και που επισκέφθηκε πέρυσι το Καζακστάν, καθώς και Ειδικό εκπρόσωπο τη Ένωση ε, ε, τονίζουν ότι τα δικαιώματα, τα πολιτικά δεν θεωρούνται ω δικαιώματα αλλά ω προνόμια. Επίσης μπορούσαμε να το απαγορεύεται η ελευθερία λόγου, συγκέντρωσης, έκφρασης κτλ. Ε, η εθνική ασφάλεια, δημόσια τάξη κυριαρχούν σε σχέση με τις ατομικές ελευθερίες δεν ε, θεωρούνται αυτά αναγκαία όπως σε μια δημοκρατική κοινωνία. Νέα ποινική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στο Καζακστάν πέρσι τον Ιούλιο και που άρχισε να ισχύει από την 1η Πρώτου φέτος αυξάνει τις ποινές κατά όσων συγκεντρώνονται σε διαδηλώσεις. Η δυσφήμιση επίσης είναι ποινικό αδίκημα. ηγέτης κάποιες δημόσιες ένωσης δεν ε, προβλέπεται να είσαι. Ε, πρόσφατα ε, ο νόμος ε, περί της προστασίας των παιδιών εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο αλλά δεν έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο. Σύμφωνα με αυτή την νομοθεσία οι πληροφορίες για το LGBT είναι βλαβεροί και απαγορεύεται. Το ίδιο πρόκειται να γίνει στο Κυργιστάν και στο Τατζικιστάν. Τώρα, σε σχέση με τους αλλοδαπούς ε, δεν έχουμε και τους πράκτορες ε, θα υποβληθεί η σχετική νομοθεσία τον επόμενο Ιούλιο, όπως προβλέπετε. Σύμφωνα με την νομοθεσία μας, όλη η, κάθε, κάθε συμβολή, κάθε έμβασμα που γίνεται πρέπει να καταγράφεται στο σχετικό μετρό στο Υπουργείο Οικονομίας. Και προτίθεται η κυβέρνηση να περάσει έναν, ε, έναν νόμο για τους ξένους πράκτορες όπως στη Ρωσία. Στο Κυριζιστάν η κατάσταση επιδεινώνεται με ραβαίους ρυθμούς και μετά από 8 χρόνια επισκέφθηκα την περασμένη εβδομάδα την πρωτεύουσα της χώρας και με εξέπληξε ότι καταγραφόταν οι συνομιλίες μου με δύο ακτιβιστές από δύο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί υπόκειται σε πιέσεις και μάλιστα Κάποιοι άλλοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη, επειδή είναι ε, ακτιβιστές. Στο Τουρκμενιστάν τέτοιες ελευθερίες δεν υπάρχουν καν. Πολλοί έχουν αυτοεξοριστεί ε, υποστηριχτές ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι ακτιβιστές. Και αυτό έχει, παρότι το Τουρκμενιστάν ανήκει στην ΟΑΣΕ, οι περισσότεροι πολιτικοί ε, αντίπαλοι του καθεστώτος είναι είτε στη φυλακή είτε στην εξορία και δεν υπάρχει ελευθερία στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Για το Καζακστάν τώρα να σας πω και κάποια θετικά στοιχεία. Πρόσφατα επικυρώθηκε η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες και η κυβέρνηση είναι τώρα πιο ανοιχτή για διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και αυτός ο διάλογος έχει θεσμοθετηθεί κάπως περισσότερο. Πρακτικά όλες οι μεγαλύτερες ε, ε, ενώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο ε, και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αυτό το οποίο ασχολείται με τον διάλογο αυτό. Θα πρέπει να σας αναφέρω τον Βλαδίμιρ Κασλόφ, που είναι, τον, τον Βλαδιμίρ Κουράμσοφ, που είναι υποστηριχτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και άλλους ακτιβιστές, οι οποίοι έχουν ε, φυλακιστεί και καλούμε την απελευθέρωσή τους, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολιτικοί κρατούμενοι για την επικείμενη συμφωνία με το Καζακστάν. Πιστεύουμε πως είναι καιρός τώρα να θίξουμε αυτό το θέμα για αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρονται πολλές φορές στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης θα πρέπει να κληθεί η κυβέρνηση του Καζακστάν να αναθεωρήσει τις πρακτικές για την επιβολή της νομοθεσίας. Έχουν και να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και να ακολουθήσει τις συστάσεις ε, το ΟΗΕ και των διαφόρων επιτροπών του. καθώς και τις απόψεις και τις εκθέσεις των ε, εκπροσώπων του ΟΗΕ που επισκέφθηκαν το χώρα πριν, εδώ και δύο χρόνια. Τώρα να σας πω και δύο λόγια για τη Ρωσία και την Ουκρανία και τις σχέσεις του Καζακστάν με τη Ρωσία. Βασικά το Καζακστάν είναι υπό την προπαγάνδα της Ρωσίας, προωθεί διάφορες θεωρίες συνομασίας και απαξιώνει τη δημοκρατία και τις δημοκρατικές αξίες. Είναι πολύ αρνητικός αντίκτυπος αυτής της προπαγάνδας στην κοινωνία του Καζακστάν. 80% των πολιτών υποστηρίζουν τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Επιπλέον ε, ανησυχεί πολύ κυβέρνηση λοιπόν ε, γίνουν τα ίδια, γιατί έχουμε μεγάλο ρωσικό πληθυσμό στη, ειδικά στα βόρεια της χώρας μας. Αυτή η ρωσική πολιτική είναι απειλή για την ανάπτυξη της χώρας και πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ελπίζω πως η συζήτηση γύρω από την ε, συμφωνία αυτή θα μπορέσει να συμβάλλει θετικά στις εξελίξεις για τη χώρα μας, αλλά και για ολόκληρη την ε, περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ε, Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τάγεβα, που είναι από το Ουσμπεκιστάν, υπερασπίζεται εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι η πρόεδρος της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κεντρική Ασία. Έχει λάβει πολιτικό άσυλο στην ε, Γαλλία και θα μας μιλήσει για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, όπως επίσης και για το δικαστικό σύστημα. Χρειάστηκε να φύγει από τη χώρα της εσπεσμένα ε, και γι' αυτό νομίζω ότι η προσωπική της ε, ιστορία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους εδώ στην αίθουσα και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο τι γίνεται στο Ουσμπεκιστάν με τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν γιορτάσουμε τα 10 χρόνια τραγωδία στην Είχαμε εκεί μια, μαζική δολοφονίας ε, της 13 Μαΐου του 2005 από τον πρόεδρο ε, κύριο Καρίμοφ και αυτή τη δεκαετία, αυτή την επέτειο ε, γιορτάζουμε σήμερα. Δυστυχώς η κατάσταση παραμένει η ίδια. Αυτή τη στιγμή το γεγονός πως έχουμε τόσα θύματα αποδίδεται στο γεγονός πως χρησιμοποιήθηκαν όπλα χωρίς προσοχή και πρέπει να σας πω πως τα όσα κάνει ο κύριος Καρίμοφ δεν επιτρέπει στο να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα της αρχές της τάξης στο Ουσμπεκιστάν. Μετά από την τραγωδία αυτή πρέπει να σας πω πως εστάλθηκε ένα μήνυμα από το Ουσμπεκιστάν εκείνη τη στιγμή ε, Συγγνώμη. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή την τραγωδία επέβαλε κάποιες κυρώσεις που έδειξαν πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ σοβαρά αυτά τα γεγονότα. Παρ' όλα αυτά οι κυρώσεις τελικά δεν εφαρμόστηκαν και ε, ξεκίνησε από εκείνη τη στιγμή και μετά μια πολιτική ανταλλαγή και να σας πω πως τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτή τη στιγμή μόνο χειροτερεύουν στο Ουσμπεκιστάν. Έχουμε χιλιάδες κρατουμένους, εκ των οποίων οι 19.000 είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Και έχουμε και 40 ε, από αυτούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα γνωστοί για τη δράση τους ε, στην κοινωνία των πολιτών. Έχουμε ε, δημοσιογράφους, αντιδραστικούς, ε, ακτιβιστές, εχθρούς του καθεστώτος. Έχουμε πάρα πολλούς. Τον κύριο Χαλτάροφ, τον ε, Νασίμ και άλλους πολλούς ακόμα. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο για ένα πρώην για τον Μουράτ Τζουράεφ, ο οποίος ε, βρίσκεται ε, ήδη 21 χρόνια φυλακή. Ξέρετε πως όταν καταδικάστηκε ζητήθηκε να μπορέσει να υποβάλει έφεση, αλλά δεν έγινε αυτό δεχτό δεκτό από την κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν. Για τα τελευταία δέκα χρόνια στο Ουσμπεκιστάν ε, κατηγορήθηκαν ε, γύρω στους 500 ακτιβιστές και διώχθηκαν και οι οικογένειές τους. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο στη χώρα. Χίλιοι ε, από τους πολίτες του Ουσμπεκιστάν αυτή τη στιγμή διώκονται καταζητούνται από την Ιντερπόλ. Ε, και ε, μέσα σε αυτούς έχουμε μάρτυρες από την τραγωδία του Ντιτζέγκ όπως επίσης ε, πολύ γνωστά άτομα τα οποία προσπάθησαν να υπερασπιστούν τους μάρτυρες αυτής της τραγωδίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε τις σχέσεις με το Ουσμπεκιστέν και αν πιέζουμε το Ουσμπεκιστάν για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτό θα οδηγήσει μόνο σε, περισσότερες, ε, σε πρόσφυγες, σε περισσότερες καταδίκες και σε μεγαλύτερη ε, πίεση επιτόπου. Εσείς δεν γνωρίζετε αυτή τη στιγμή πως για παράδειγμα το δικαίωμα της ιδιοκτησίας δεν γίνεται σεβαστό ε, στο Ουσμπεκιστάν. Η η εφορία είναι πάρα πολύ ε, διεφθαρμένη. Ο Μπατήρ Παρπίφ που είναι ε, κοντινός συγγενής ε, του αρχηγού της ε, υπηρεσίας πληροφοριών αυτή τη στιγμή έχει πλουτίσει και παρόλο που είναι από τους ανθρώπους για τους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή βασιλεύει. Κανείς, κανείς αρχηγός κράτους ε, με συγχωρείτε, κανένα από όσου ήταν στην ηγεσία τη χώρα μα τα τελευταία 26 χρόνια δεν έχει υποβάλει πόθεν έσχε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε αυτή την κατάσταση να ε, εξασφαλίσουμε μια ε, δίκαιη δίκη και να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή. Οι επιχειρηματίε του Ουσμπεκιστάν γίνονται πρόσφυγε. Ζητούν το δικαίωμα να να χαρακτηριστούν ως πρόσφυγες και παρόλα αυτά μετά από ορισμένου μήνες τους επιστρέφουν στη χώρα όπου έχουμε προβλήματα με την ε, δωροδοκία, με τη διαφθορά. Ε, πολύ συχνά οι μεταναστευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν λαμβάνουν υπόψη το γεγονός πως οι άνθρωποι με την Κεντρική Ασία δεν μπορούν να αποδείξουν πως το γεγονός πως διώκονται έχει να κάνει με τα πολιτικά τους πιστεύω και πολλές φορές να σας δώσω ένα παράδειγμα το 2014 ο Βαχραντίν Τελάιφ ο οποίος ήταν ε, ε, κρατούμενος βασανίστηκε. Ζητήκε ο συνήγορός του να γίνει μια ετροδικαστική εξέταση και το δικαστήριο δεν έδωσε αυτό το δικαίωμα. Για τα τελευταία δέκα χρόνια η Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κεντρική είπε πως έχουμε 114 δολοφονίες, απαγωγές, βασανισμούς, όσων από τους, ε, από, ε, από τους ολιγάρχες στη χώρα μας, από τις αρχές, όπως επίσης ε, και από ε, ε, μέλη της κυβέρνησης. Για αυτούς που είναι από το Καραπακαλστά να σας πω πως ζουν μέσα σε ένα πολύ δύσκολο, δύσκολο περιβάλλον. Κανείς όμως δεν τους θεωρεί ότι είναι πρόσφυγες λόγω περιβαλλοντολογικών δυσκολιών παρόλο που η χώρα τους έχει, έχει καταστραφεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ζητήσει και πάλι αυτά τα οποία ζητούσε από τους Πακιστάν το 2009 πριν άρει τις κυρώσεις και μέχρι σήμερα αυτά δεν γίνονται σεβαστά. Όπως επίσης το ψήφισμα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2014. Θα πρέπει εσείς να επενθυμίσετε για μια φορά ακόμα στο Ουσμπεκιστάν που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, εφαρμόσει αυτό το ψήφισμα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει όλα αυτά τα πολιτικά στοιχεία υπόψη. Η Ένωση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, Κεντρική Ασία ε, και η Human Rights Watch, όπως επίσης και η Amnesty International, η FEDEAS. Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις οι οποίες απευθύνουν μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τις χώρες αυτές να επιτρέψουν μία ανεξάρτητη επιτροπή να διερευνήσει τα αίτια της ε, τραγωδίας ε, στη χώρα. έχουν εξαφανιστεί δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, όλα αυτά θα πρέπει η Human Rights Watch στα συμπεράσματα που βγάζει να ακουστεί. Χρειάζεται διεθνής βοήθεια για το Ουσμπεκιστάν. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε πώς μπορούμε ε, ο Ερυθρός Σταυρός, για παράδειγμα, να ξαναλειτουργήσει στη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό το Ουσμπεκιστάν να έχει... Ε, εκεί να έχει πρόσβαση ο ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ, ο οποίο εδώ και 10 χρόνια δεν επιτρέπεται να επισκεφθεί τη χώρα. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση του Ουσβεκιστάν δεν δέχεται να συνεργαστεί ε, με τον ΟΗΕ, και που παραβιάζει ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου ε, συνέχεια, θα πρέπει να απευθυνθούμε να απευθυνθούμε στον ειδικό εισηγητή για το Ουσμπεκιστάν και να ζητήσουμε να εφαρμοστούν κάποιες κυρώσεις. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την τραγωδία στην Τιτζάν και θα ήθελα να βασίζομαι στη νέα στρατηγική που θα ακολουθήσετε εσείς για τις σχέσεις με το Ουσμπεκιστάν. Εγώ είμαι πολίτης του Ουσμπεκιστάν και θα ήθελα στη δική μου χώρα το δικαίωμα του, της του λόγου να γίνεται ε, σεβαστό, να υπάρχει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, να μπορούμε να, σεβαστούμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει μια ιστορική ευκαιρία να φέρει την αλλαγή και να προωθήσει τη δημοκρατία στο Ουσμπεκιστάν. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα συνεχίσουμε με αυτή τη σειρά. Η κυρία Μαρία Ρένα βρίσκεται εδώ και επειδή θα συζητήσουμε για το ίδιο κράτος που είναι το Ουσμπεκιστάν, μια και η ίδια είναι η ειδική εισηγήτρια για τα κλωστιφαντουργικά που συνδέονται με την Συμφωνία Εταιρική Σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Θα ήθελα τώρα να τη δώσω το λόγο. Κυρία Ρένα. Και μετά θα συνεχίσουμε. Bienvenida. Merci, euh, Madame la Présidente. Merci, Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Έλενα. Είναι αλήθεια ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτήν την Επιτροπή ε, και είναι μεγάλη μου η χαρά, καθώς επιπλέον ε, συχνά μας λένε ότι η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα μέσο που έχει στη διάθεσή της και που είναι σημαντικό και είναι αυτό οι συμφωνίες ε, εμπορικής εταιρικής σχέσης για να μπορέσει δηλαδή να επηρεάσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους. Είναι λοιπόν ε, μεγάλη μου χαρά που μπορούμε να αναλύσουμε την κατάσταση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, την ΙΝΤΑ, και ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία, αυτό το πρωτόκολλο για την κλωστή παντουργία το οποίο το διαπραγματευτεί και ε, ανάμεσα στην Κομισιόν και τις αρχές του Ουσμπεκιστάν και σήμερα αυτό το πρωτόκολλο είναι σε αναμονή. Ε, κάποιες συστάσεις είχαν διατυπωθεί από το κοινοβούλιο μας ε, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του θέματος της κλωστηθαντουργίας και ιδιαίτερα στο θέμα της εργασίας των παιδιών στη συλλογή του βαμβακιού αλλά και σε όσα έχουν να κάνουν με το θέμα της Σε Σήμερα αυτό το πρωτόκολλο είναι πάλι στην ημερήσια διάταξη. Ζητήσαμε να γίνουν ιδιαίτερα ακροάσεις και να μας δοθούν υποδείξεις από, από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για να δούμε αν οι συστάσεις που είχαν διατυπωθεί τότε έχουν βρει ανταπόκριση. Ορισμένε πληροφορίες μας δόθηκαν από διάφορες οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλο ιδιαίτερω όσον αφορά το δικαίωμα ε, στην εργασία για τα παιδιά, ότι ίσως θα είχαν ε, υπάρξει κάποιες βελτιώσεις, αλλά ότι ταυτόχρονα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία. Αλλά αυτό αφορά τους ενήλικες καθώς και ότι πρόκειται για μια κρατική πρακτική όσον αφορά την καταναγκαστική εργασία. Αύριο θα γίνει η ακρόαση όσον αφορά την ε, συγκεκριμένη κατάσταση της εργασίας της παιδικής εργασίας αλλά και της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουσμπεκιστάν, πράγμα που ίσως θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την εντολή που δόθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για να δουλέψει για αυτή την κατάσταση στα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργατικά δικαιώματα στο Ουσμπεκιστάν και τη βάση αυτής της ανάλυσης θα ε, λάβει θέση το Κοινοβούλιο. Μετά από τις ακροάσεις δηλαδή που θα έχουν γίνει με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρω πως η κατάσταση δεν είναι απλή ούτε για εκείνους στο Ουσμπεκιστάν για να κάνουν την ανάλυση και να μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε λοιπόν τέτοια μέσα όπως οι εμπορικές συμφωνίες ώστε η Ευρώπη να παίξει καταλητικό ρόλο ε, στις αλλαγές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες. Θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση. Θα ήθελα να σε εξηγήσω ποια είναι η δική μας προσέγγιση και να σα πω πως δυστυχώς το Ουσμπεκιστάν αυτή τη στιγμή επειδή ακριβώς έχουμε αυτή τη μαζική εκμετάλλευση είναι πολύ ψηλή η θλισιμότητα. Κανείς στην πραγματικότητα δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το θέμα. Τα, τα θύματα τα οποία τραυματίζονται ακριβώς λόγω αυτής της καταναγκαστικής εργασίας, οι συγγενείς που χάνουν τα παιδιά τους, όπως επίσης και αυτοί που ζουν κοντά σε αυτά τα χωράφια, φοβούνται και όλα αυτά τα επεισόδια ε, αποσιωπώνται και ελέγχονται βεβαίως πάντα οι πληροφορίες που γίνουν από τις υπηρεσίες πληροφοριών και δεν έχουν και το δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να βγουν από τη χώρα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούμε να μελετήσουμε αυτό το θέμα της μοντέρνας δουλείας στο Ουσβεκιστάν. και εσείς είδατε πως αυτή υπάρχει, υπάρχει, υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες καταγγελίες και είδαμε ποιες ήταν οι αποφάσεις των δικαστηρίων οι οποίοι ε, θεωρούν πως πρόκειται μία από τις υποχρεώσεις που έχει ο πολίτης προς την κυβέρνησή του. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαρία, θέλεις κάτι ακόμα. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συζήτηση. Νομίζω πως εδώ Έχουμε τον ΤΕΣ και το Ουσμπεκιστάν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έτσι ώστε να είναι πιο πλήρης οι πληροφορίες που έχουμε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γιούρι Τζιμπλάτζε από το Κέντρο για την Ανάπτυξη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Μόσχα. Είναι λοιπόν η βάση του στην ε, Ρωσία και θα μας κάνει μία περιγραφή της κατάστασης των ανθρώπων ανθρώπινων δικαιωμάτων σε κάποια κράτη και εδώ θα συμπεριλάβουμε και το Τουρκμενιστάν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Εγώ μιλώ εξ ονόματος της εξαιρετίας αποδείξεις ότι ζουν. Ε, μια εκστρατεία που ξεκίνησε το 2013 από ένα συνασπισμό ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από ευρωπαϊκές χώρες στην Βόρεια Αμερική αλλά και ακτιβιστές εντός του Τουρκμενιστάν με στόχο να προστατευτούν τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους καθώς και να καταγγείλουμε την πρακτική των καταναγκαστικών εξαφανίσεων στο Τουρκμενιστάν. Φυσικά αυτή η συζήτηση η σημερινή δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη το να ασχοληθούμε με την ανθρώπινη κατάσταση στο Τουρκμενιστάν και να εξετάσουμε τι δυνατότητε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επηρεάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου σε αυτή τη χώρα είναι απόλυτα απαραίτητο στη στιγμή που το επίπεδο ε, της αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα, ε, ανάμεσα στα δύο μέρη μάλλον ε, και οι συνομιλίε έχουν φτάσει σε νέα εξέλιξη. Η κύρωση της ε, συμφωνίας είναι και πάρα στην ατζέντα του Κοινοβουλίου και προχωρά γρήγορα και προγραμματίζεται η κύρωση στις επόμενες εβδομάδες, ενώ ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσεις με τις τουρκμενικές αρχές για την κατασκευή του αγωγού ε, μέσω της ε, Κασπίας ε, έχουν φτάσει επίση επίσης σε νέο στάδιο. Ήδη έχουν γίνει μελέτες ε, και περιβαλλοντικές μελέτες. Στη διάρκεια της επίσκεψης στο Άσχαμπατ την περασμένη εβδομάδα, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σεύκοβιτσα ανακοίνωσε ένα σχέδιο ώστε να εξασφαλιστεί η πρώτη παράδοση του τουρκμενικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη το 2019, πολύ σύντομα δηλαδή επιπλέον των ισχυρών αμοιβαίων ε, συμφερόντων ε, για την αγωγούς φυσικού αερίου, η κρίση στην ε, Κρυμαία οδηγεί το Τουρκμενιστάν να προβεί και την Ένωση να προβεί σε γρήγορη ολοκλήρωση αυτή τη συμφωνία με το Τουρκμενιστάν είναι η μόνη χώρα τη Κεντρική Αφρική, Ασίας, με που δεν έχει τέτοιου είδου συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διαδικασία προετοιμασία μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση του Τουρκμενιστάν. Πριν από πέντε χρόνια είχε γίνει, είχε απορριφθεί τέτοια συμφωνία λόγω τη παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά τη τουρκμενική κυβέρνηση και είχαν προταθεί διάφορα ορόσημα στι εκθέσει και τα ψηφίσματα που έγιναν από το 2006 μέχρι και το 2010. Φυσικά υπάρχουν πολλά περισσότερα από ό,τι απλά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχέση μεταξύ Ένωση και Τουρκμενιστάν και τα στρατηγικά συμφέροντα για την ενέργεια τη ε, Ένωση πρέπει πολύ σοβαρά να ληφθούν υπόψη. Ωστόσο, πρέπει να δούμε τι έχει γίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα από το 2010 η κατάσταση παραμένει μία από τις χειρότερες στον κόσμο και τα τελευταία πέντε χρόνια δεν φαίνεται να έγιναν σημαντικές βελτιώσεις σε όλους τους τομείς όπου έπρεπε να δοθεί ε, πηγόντως προσοχή. Βασικά όλα τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα και ελευθερίες ε, παραβιάζονται κατάφορα ή λείπουν, εκλείπουν τελείως οι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές, ακόμα και αυτοί που ζουν στην εξορία, αντιμετωπίζουν διαρκώς απειλή ε, βίαιης καταστολής από την κυβέρνηση. Ε, τα, λεπτά ζητήματα μπορούν μόνο κρυφά ή στην εξορία να ε, συζητηθούν. Οι δημόσιες συγκεντρώσεις είναι σπάνιες γιατί υπάρχει φόβος ε, για, όσον αφορά την επίκριση οποιασδήποτε επίσημης κρατικής πολιτικής. ο, το κράτος ελέγχει τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ε, ε, και τα κοινωνικά δίκτυα καθώς και πολλά sites είναι μπλοκαρισμένα. Πλήρης, απόλυτος και διαιτητικός ε, κυβερνητικός έλεγχος απεδείχθηκε πρόσφατα μέσω της κυβερνητικής εκστρατείας ώστε να ε, καταρρύψει όλους τους δορυφόρους που μποροσέφεραν ανεξάρτητη ενημέρωση στο κοινό του Τουρκμενιστάν. Διεθνείς, ε, εκπομπέ εκπομπές από διεθνή κανάλια δεν επιτρέπονται. Επίσης, δεν μπορεί ο κόσμος να ταξιδέψει. Γίνονται απλώς αυθαίρετες απαγορές απαγορεύσεις ε, μετακίνησης. Ε, τέτοιες απαγορεύσεις μπορεί επίσης να επιβληθούν στον οποιονδήποτε, όχι μόνο σε ακτιβιστές ή αντικυβερνητικούς και τις οικογένειές τους, αλλά και σε φοιτητές. Βασανιστήρια επίσης είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτό αντικατοπτρίζει την, ε, την ιδιαίτερα αυθαίρετη ε, φύση του συστήματος. Συστηματικά χρησιμοποιούνται για την δίωξη των αντιφρονούντων. βασανιστήρια γίνονται στην περίφημη ε, φυλακή ε, που είναι η φυλακή, η φυλακή του Οβαντάν Τεπέ ή πιο γνωστή φυλακή για τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια που γίνονται εκεί. Ξεχωρίζει το Τουρκμενιστάν από όλους τους γειτονές του που είναι επίσης ε, αυταρχικά και καθεστώτα. Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί από τις τουρκμενικές φυλακές και έχουμε τα τεκμήρια στις εκθέσεις μας. Ε, άλλες εξαφανίσεις ε, ε, γίνονται και στην Τσετσενία, στην πρώην Κοσλαβία, στην Ανατολική Ουκρανία, όμως εδώ πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό εξαφανιστέντων σε μια χώρα στην Ευρωασιατική περιοχή. Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων ήταν αυτοί που υποτίθεται ότι προ... σχεδίαζαν την δολοφονία του Προέδρου του Τουρκμενιστάν, του Σαμπαραμουράτ Νιγιάζοφ, το 2002. Αν και άλλοι έχουν καταδικαστεί για μη πολιτικά εγκλήματα σε διάφορα κύματα καταστολής. Ε, ε, ε, οι περισσότεροι βρίσκονται στη φυλακή χωρί κανεί να ξέρει τι του συμβαίνει. Περισσότεροι για 12 χρόνια. Και τελευταία φορά που του είδε κανεί ήταν όταν συνελήφθησαν οι δε αποδείξεις που έχουμε συλλέξει από την εξαρτία μας ε, λένε, τα στοιχεία μάλλον που έχουμε συλλέξει, δείχνουν ότι όλοι αυτοί έχουν υποστεί βασανιστήρια και πολύ κακή μεταχείριση. Υπάρχουν επίσης μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι ορισμένοι έχουν πεθάνει στις φυλακές. Ορισμένοι ε, φυλακισμένοι, ε, κρατούμενοι, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να απελευθερωθούν το 2003-2014 καθώς θα είχαν κτίσει την ποινή τους, όμως ε, οι συγγενείς τους έμαθαν από τις αρχές ότι νέα ε, ποινή τους είχε ε, επιβληθεί χωρίς καμία δικαιολογία. Σε κάποιες φορές υπό τη μορφή συλλογική τιμωρίας οι οικογένειες των εξαφανιστέντων συνελήφθησαν ή απολύθηκαν από τις δουλειές τους, ε, κατασχέθηκαν ε, οι περιουσίες τους και πολύ συχνά ε, τους απαγορεύθηκε να ταξιδέψουν. Αυτές οι πολιτικές ε, καταστολές, τα βασανιστήρια, οι συνοπτικές δίκες καθώς και οι εξαφανίσεις ε, στο Τουρκμενιστάν ήταν η ε, αντικείμενο διεθνούς ανησυχίες. Από το 2013 έχουν γίνει ψηφίσματα του Συμβουλίου του ΟΗΕ και δηλώσεις της ΟΑΣΕ. Ωστόσο, η πρακτική των ε, εξαφανίσεων συνεχίζεται υπό τον ε, πρόεδρο Μπέρντι Μουχαμέτοφ, αν και σε μικρότερη κλίμακα. Γνωρίζουμε τουλάχιστον 7 τέτοιες περιπτώσεις. Η χώρα είναι κλειστή. Δεν Κανένας ανεξάρτητος οργανισμός δεν έχει μπει για να δει τι συμβαίνει. Οι ε, αντίστοιχες τα, τα, τα αιτήματά μας που γίνονται εδώ και καιρό δεν έχουν καν λάβει απάντηση. Διάφοροι νέοι νόμοι συμπεριλαμβανομένου του νόμου για την ε, ελευθερία συγκέντρωσης και για το ελεύθερο, ελεύθερο ίντερνετ ε, ε, υποδεικνύονται από την κυβέρνηση ως πρόοδος, γιατί η κυβέρνηση θέλει να κάνει ότι προοδεύει. Ωστόσο, αυτές οι νέες νομοθεσίες ε, ακολουθούν μια πολύ περιοριστική προσέγγιση και είναι πιθανό να καταλήξουν σε οποιαδήποτε πραγματική βελτίωση αν δεν ληφθούν σοβαρά και συστηματικά μέτρα για να θεσπιστεί μια πιο δίκαιη ε, κοινωνία. Συνταγματική μεταρρύθμιση δε που υποτίθεται ότι θα γίνει δεν θα επεκτείνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερία Ωστόσο πιστεύουμε πω αυτή τη στιγμή έχει προκύψει πριν από λίγους μήνες μια μοναδική ευκαιρία ώστε να πιέσουμε για πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα και για του εξαφανιστέ του Τουρκμενιστάν χάρη στο συνδυασμό πολιτικών και νομικών παραγόντων. Το πρώτο σύνολο παραγόντων είναι η άνευ προθυμία των ε, τουρκμενικών αρχών να αναπτύξουν σχέσεις και να αρχίσουν ε, ενεργή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη δυτική κοινότητα λόγω των οικονομικών και ε, αναγκών που είναι μία ε, ανάγκη πολύ έντονη. Τώρα πολλά ε, φυσικό αέριο το Τουρκμενιστάν στην Κίνα, αλλά πολύ πιο φτηνό και σε πολύ μικρότερους όγκους από το παρελθόν, οπότε, μας ε, οπότε λείπουν έσοδα. Χρειάζεται διαφοροποίηση, τεχνολογία, υποδομές. Το Τουρκμενιστάν αυτά δεν τα έχει. Ενώ η Ένωση ενδιαφέρεται να εισάγει φυσικό αέριο από το Τουρκμενιστάν ώστε να διαφοροποιήσει τις ε, πηγές ε, ενέργειας και να ξεφύγει από το μονοπόλιο της Γκασπρόμ και της Ρωσίας. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ανάγκες αυτές του Τουρκμενιστάν ε, να πουλήσει φυσικό αέριο στην, φυσικό αέριο στην Ένωση ώστε να πιέσει για βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα. η κυριαρχία της Γκάσπρομ έχει χτυπήσει το Τουρκμενιστάν. Έχουν μειωθεί τα αποθέματα και το Τουρκμενιστάν χρειάστηκε να εγκαταλείψει την ε, δωρεάν παροχή βασικών αγαθών όπως ε, τα αγαθά και υπηρεσίες προς τον πληθυσμό. Πράγμα το οποίο χρησιμεύσε ως θεμέλιο για το κράτος προνοίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, Απειλή ασφάλειας από το Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν οργανώνουν επιθέσεις ε, το 2014 και το 2015 πολύ κοντά στα σύνορα με τη χώρα του Τουρκμενιστάν με θύματα ε, ε, Υπάρχουν αναφορές για αυξανόμενη παρουσία ε, σωμάτων του Ισλαμικού κράτους ανησυχούν το Τουρκμενιστάν πάρα πολύ και το πιέζουν για στενότερες σχέσεις με τον έξω κόσμο ε, για λόγους ασφάλειας και δεν επιλέγουν τη Ρωσία αλλά την Δύση λόγω του ότι φοβούνται την επιθετική πολιτική της Ρωσίας ε, από πέρυσι. Αυτές οι ανάγκες λοιπόν για, για επαφή με την ε, έξω κόσμο δίνουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ ε, καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Βέβαια, οι τουρκμανικές αρχές θέλουν να έχουν σχέσεις με το διεθνή κοινότητα, χωρίς όμως να κάνουν αλλαγές. Τώρα, νομική ε, ε, είναι οι λόγοι επίσης ε, συμπεριλαμβανομένου της 20ης επαιτίου του καθεστώτος ουδετερότητας, επίσης υπεροχή των διεθνών κανόνων σε σχέση με την χώρια νομοθεσία και η πρόσφατη αναθεώρηση του ποινικού κώδικα προβλέπει την αναδρομική εφαρμογή, δηλαδή διάφοροι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για πολύ χρόνο θα έπρεπε ήδη να έχουν απελευθερωθεί, αλλά αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Στο πλαίσιο του UPR το 2013 το Τουρκμενιστάν υιοθέτησε διάφορες συστάσεις άμεσα συνδεδεμένες με τα βασανιστήρια και τις συνθήκες της κράτησης και δεσμεύτηκε να βελτιώσει ε, τις συνθήκες κράτησης των κρατουμένων που ε, εκτίων πολύ μακροχρόνιες ποινές και μόλις πριν από λίγους μήνες υιοθέτησε μια πολύ σημαδιακή ε, απόφαση για ένα μεμονωμένο, μια μεμονωμένη καταγγελία όπου αναγνωρίζει τον χώρο της Μουράνταφ, που είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους εξαφανιστέντες, πρώην υπουργό του Τουρκμενιστάν και ε, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ως θύμα αναγκαστικής εξαφάνισης και η σύζυγός του επίσης έπεσε θύμα βασανιστήριων ε, και αναγνωρίστηκε. Πρόκειται για τον Μπόρις Σιγκμουράτοφ. Φαίνεται λοιπόν ότι ε, η επιθυμία για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ ε, ισχυρό εργαλείο για αυτήν. Ε, Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Μία κύρωση της συμφωνίας μπορεί να εξαρτάται από τα ανθρώπινα δικαιώματα ή από νέους δρόμους ε, προόδου μετά την ε, κύρωση έτσι ώστε να υπάρχει ένας τρόπος ε, να αναφερόμαστε στα θέματα αυτά με προς την κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν. Δηλαδή ένα είδος μοχλού που θα μας επιτρέψει αφού επικυρωθεί η συμφωνία αυτή να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτό που προτείνουμε είναι η κύρωση της συμφωνίας να εξαρτηθεί από πραγματική πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα που ακόμα δεν έχει λάβει χώρα. Ακόμα δεν έχουμε καθόλου πρόοδο σε σχέση με πέντε χρόνια και τα θέματα που είχατε θίξει εσείς τότε εξακολουθούν να, να παραμένουν ενισχύ και μάλιστα το σημείο αναφοράς για τις συγκρίσεις θα πρέπει να παραμείνει εκεί που βρίσκεται. Η κύρωση λοιπόν ε, της συμφωνίας είναι πολύ σημαντική για το Τουρκμενιστάν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σε μια μοναδική θέση για να πιέσει αυτά τα, τα αιτήματα και να θέσει την πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα ως κομβικό σημείο για την υπογραφή και την κύρωση της συμφωνία, Την κύρωση, με της συμφωνίας διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών για να δούμε ποιοι θα είναι οι δείκτες αναφοράς και μέχρι στιγμής υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος ε, ρεαλιστικών ετοιμάτων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μέσα σε μία περίοδο κάποιων μηνών. Δεν συμφωνούμε με το επιχείρημα που λέει πως η κύρωση ε, της συμφωνίας ε, θα είναι αποτελεσματική από μόνη της, γιατί θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την τουρκμενική κυβέρνηση και αυτό θα γίνει μέσω της ενδεχόμενης επικύρωσης που θα λάβει η χώρα εάν κάνουν κάποια βήματα πρόοδο. Είναι λοιπόν δύσκολη αυτή η στιγμή γιατί έχουμε τους σκληρούς στην κυβέρνηση της χώρας που θέλουν να δοκιμάσουν τα όρια μας και να δουν αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβιβαστεί και να υπαναχωρήσει σε σχέση με τις προηγούμενες θέσεις της. Εάν λειτουργήσει τότε θα καταλήξουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδύναμη και μπορεί να χειραγωγηθεί και για άλλα θέματα, ίσως και εμπορικά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αυτή η σπουδή. Γιατί δηλαδή υπάρχει εδώ το χρονοδιάγραμμα για την ακύρωση και χρειάζονται μόλις τρεις μήνες μετά από αυτή τη μακρά περίοδο αναστολής και από τη στιγμή που δεν ε, έχει χρησιμοποιηθεί η κύρωση ως μοχλός πίεσης. Εμείς λέμε ότι καλό θα ήταν να αναβάλλετε εσείς τη συγκατάθεσή σας στην κύρωση. Να πείτε πως θα εξαρτηθεί από μετρήσιμού δείκτες αναφοράς, θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πως σε έξι μήνες ή ένα χρόνο θα ξαναεξετάσετε το θέμα. Χρειάζεται ένας μηχανισμός παρακολούθησης στεναρός που θα μπορούσε να είτε ε, από τη δική σας υποεπιτροπή, είτε από την ΑΦΕΤ, είτε από τον ειδικό εισηγητή, είτε από τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα βοηθήσουν εκεί και οι μη καπαόμικρον. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο ε, μηχανισμός επιτήρησης θα υποσκάψει αυτό το γεγονό στην θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ε, γενικότερη ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα τους εκπροσώπους της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης που μπορούν αυτή τη στιγμή να απαντήσουν σε ένα μεγάλο κομμάτι από τις ανησυχίες που ακούστηκαν. και σίγουρα ε, όλοι στην Επιτροπή μας έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Είστε πολλοί. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ο κύριος Γκάριθ Ομπράιεν που είναι ο policy officer για τη στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρμογή αυτών ή θέλετε να ξεκινήσει κάποιος άλλος. Θέλετε να τα πείτε χώρα-χώρα. Εσείς ε, αποφασίστε. Κύριε Γκάριθ Ομπράιεν πάρτε το λόγο αν θέλετε. Θα ξεκινήσω εγώ. εγώ. Το είμαι υπεύθυνο της, ε, του τμήματος Κεντρικής Ασίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Συμφωνώ με του ομιλητές πως υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην ε, Κεντρική Ασία και πράγματι είχαμε κάποιες ε, θετικές εξελίξεις σε κάποιες χώρες μεταξύ των οποίων και νομοθετικές ε, μεταρρυθμίσεις, αλλά η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παραμείνει ανησυχητική στην Κεντρική Ασία. Οργανώσει των πολιτών, δημοσιογράφοι και οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν πίεση σε πολλέ χώρε ε, τη περιοχή. Υπάρχουν ε, κατασταλτικοί μηχανισμοί και παρενόχληση από την αστυνομία. Υπάρχει επίση κακομεταχείριση κρατουμένων παρά τα κάποια θετικά βήματα για την πρόληψη βασανιστήριων σε κάποιες χώρες ε, της ε, περιοχής. Ε, μειονοτικές ομάδες, θρησκευτικές μειονότητες και η κοινότητα των ΛΟΑΤ αντιμετωπίζουν διακρίσεις από το κράτος. Με την εξαίρεση της Κυργιζίας η δημοκρατία δεν έχει εδρεωθεί στην περιοχή και οι εκλογές ε, είναι είτε νόθες ε, είτε καθόλου αξιόπιστες. Η στρατηγική μας για την Κεντρική Ασία λέει πως το κράτος δικαίου, ο δημοκρατισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τη βάση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της Κεντρικής Ασίας και αυτά είναι ένα κεντρικό στοιχείο της σχέσης της Ένωσης με τις χώρες της περιοχής. Τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο φύγουμε συστηματικά στις συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αλλά θα ήθελα εδώ πέρα να τονίσω πως ε, ενώ έχουμε έναν δομημένο πολιτικό διάλογο με τέσσερις από αυτές τις χώρες, με το Τουρκμενιστάν ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, διαλόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε και με τις ε, πέντε αυτές κεντροασιατικές χώρες. Δεν συμφωνώ πως ε, οι διάλογοι αυτοί επειδή γίνονται και κλεισμένων των θυρών δεν έχουν αξία θεωρώ πως έχουν μεγάλη αξία γιατί επιτρέπουν την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και ακόμα και το να φύγουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν οδηγούν πάντα σε ουσιαστικό αποτέλεσμα αλλά έχουν οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα και βεβαίως ε, συνεχίζουμε να πιέζουμε τις ε, χώρες ε, αυτές να κάνουν περισσότερα και σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να κάνουν πολύ πολύ περισσότερα μαζί με τις ε, πρεσβείες των κρατών μελών έχουμε τακτικές συναντήσεις ε, με υπεραστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συναντόμαστε και με υπεραστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις Βρυξέλλες ε, και στις εν λόγω χώρες πριν από κάθε δημιουργή συνάντηση. Σεμινάρια επίσης που όπου συναντώνται οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και οι πανεπιστημιακοί έχουν γίνει αρκετά. Οι συστάσει αυτών των σεμιναρίων ε, για ζητήματα όπως η ελευθερία του τύπου και τα βασανιστήρια είναι κάτι το οποίο φύγουμε στους ε, διαλόγους. Στηρίζουμε εμείς ε, τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή στο πλαίσιο της ε, πρωτοβουλίας κράτους δικαίου για την Κεντρική Ασία έγινε μια σειρά σεμιναρίων για ζητήματα που είναι προτεραιότητα για όλες αυτές τις χώρες. Πρόσβαση δικαιοσύνη, αρχές ε, ε, δίκαιης δίκης, εκπαίδευση δικαστών και συνεργαζόμαστε στενά με τα γραφεία του ΟΑΣΕ, του ΟΗΕ και της υπηρεσίες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα τώρα να θίξω κάποια άλλα ζητήματα. Για το Ουσβεκιστάν βεβαίως αυτά θα τα ξαναπούμε και αύριο. Και δεν θέλω να μπω πολύ στις ε, λεπτομερίες, θα τα πω αύριο στην ε, αρμόδια επιτροπή, αλλά θεωρούμε πως μαζί με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο το στην παιδική εργασία και στην καταναγκαστική εργασία. Δεν είναι γρήγορη η πρόοδος και οπωσδήποτε δεν είναι τόσο γρήγορη όσο θα επιθυμούσαμε. Αλλά μαζί με την Παγκόσμια Τράπεζα, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, επιτυγχάνουμε κάποια πρόοδο και ελπίζουμε πως θα έχουμε ακόμη περισσότερη. Οπότε Πρόκειται για κάτι το ευρύτατο, μια ευρύτατη συνεργασία με τη συνεργασία και της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, για να μπορέσει το Ουσμπεκιστάν να απαλλαγεί από αυτά τα δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τα πράγματα προχωράνε. Για το Τουρκμενιστάν είναι δύσκολη χώρα οπωσδήποτε και δεν υποτιμούμε τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε ε, για εμάς το ερώτημα είναι αν θα επιδιώξουμε κάποια αλλαγή μέσω των επαφών ή αν θα μείνουμε στο περιθώριο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο περιθώριο. Δεν έχουμε τακτικές πολιτικές επαφές που θα μας επιτρέψουν να ασχοληθούμε με σοβαρά ζητήματα. Χωρίς δε την διάσκεψη αυτή δεν θα έχουμε τέτοιο φόρουμ ούτε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, υψηλόβαθμων αξιωματούχων, βουλευτών. Θεωρούμε λοιπόν πως η διάσκεψη αυτή είναι σημαντική για να ασχοληθούμε με κάποια από αυτά τα ζητήματα. Η αίρεσιμότητα για την κύρωση και όπως αναφέρθηκε δεν ε, έχει υπάρξει κάποιο πρόοδο σε αυτό το μέτωπο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συμφωνία αυτής της σύνδεσης δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή της διαδρομής. για η οποία θα μας επιτρέψει να δούμε με τρόπο δομημένο όλα αυτά τα ζητήματα που όλοι θεωρούμε πολύ σημαντικά. Χωρίς τη συμφωνία αυτή σύνδεση και συνεργασία δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το φόρουμ, κάτι το οποίο θα είναι λυπηρό. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους που ήρθαν να μας ακούσουν σήμερα. Και αν υπάρχει κάτι παραπάνω από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάντως που ήρθατε και για τις εξηγήσεις που δώσατε. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο πρώτος. Ίσως δεν ξέρω αν μπορούσε να μας πει κάτι περισσότερο η Κομισιόν σε σχέση με <laughs> αυτά που είπε. Καταλαβαίνω και τις δυσκολίες, διότι το να συνδυάσουμε τα συμφέροντα με τις αξίες αλλά και να έχουμε και ενεργειακή αυτάρκεια ενώ να προωθούμε τα δικαιώματα που παραβιάζονται είναι ευαίσθητη ισορροπία ε, στις σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της Κεντρικής Ασίας. Ωστόσο, είναι απόλυτα προφανές από κατά μας δεν ξέρω αν οι συνομιλητέ μα, αλλά από ό,τι κατάλαβα συμφωνούμε σε αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται κατά κάποιο τρόπο ότι τίτε στο πώ χειρίζεται χειρίζεται τα θέματα απέναντι σε αυτή τη δικτατορία του φυσικού αερίου. Ωστόσο, η ενεργειακή ασφάλεια και η πρόθεση της δημοκρατίας είναι και τα δύο κύρια σημεία της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Στην περίπτωση του Τουρκμενιστάν, θα πρέπει να σας πω ότι και εδώ υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να επιληθεί, γιατί εμείς όντως θέσαμε όρους. Όμως δεν κατέστησαν δυνατά τα ε, βήματα έμπροστα Η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάται μήπως χάσει την ενεργειακή αγορά. απέναντι στη Ρωσία και την Κίνα και δεν επιμένει ιδιαίτερα. Και ο κίνδυνο είναι να επανέλθει στην ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον τη δική μα υποεπιτροπή, να θυσιαστούν στο βωμό των οικονομικών συμφερόντων τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό για μας δεν είναι αποδεκτό. Δεν ξέρω κατά πόσο η Κομισιόν προσπαθεί να κάνει συμφωνίες που τουλάχιστον θα βάζουν στην ημερήσια διάταξη το θέμα της πρόθεσης των κοινωνικών ε, ε, προδιαγραφών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει για αυτά τα θέματα στο Τουρκμενιστάν. κάνω μια ερώτηση και μια σύντομη παρατήρηση. Καταρχήν, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο από τη δική μας πλευρά, επί τη βάση των όσων ακούσαμε, είναι απαραίτητο να ζητήσουμε να τεθεί πολύ πιο έντονα στις κατευθύνες γραμμές που ορίζονται ε, για το θέμα της κατευθύνες γραμμής στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι το πιο αδύναμο τμήμα των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει στην τελευταία φάση. Ενώ όσον αφορά το Τουρκμενιστάν, έχω μια περιέργεια για το ρόλο που, για παράδειγμα, που ασκεί το KNB. Γιατί από όσο γνωρίζω, ένα από τα στοιχεία αυτής της χώρας είναι ακριβώς αυτό που ε, θα σπάσει το φαύλο κύκλο. Η χρήση δηλαδή των υπηρεσιών να μην χρησιμοποιούνται ειδικέ υπηρεσίε για να καταργούνται στην ουσία τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προσωπικέ ελευθερίε. Θέλω να ξέρω λοιπόν ποιο ακριβώ είναι ο ρόλο του, ΚΑΠΑ, του ευχαριστω uh, πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ που ήρθαν και μας μίλησαν σήμερα για θέματα καυτά για την Κεντρική Ασία. Για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή. Και είναι πάρα πολύ απογοητευτικό αυτό το οποίο μας περιέγραψαν εδώ οι εμπειρογνώμενες στα θέματα αυτά και οι εντυπωσίε. Θεωρώ ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και ίσως δεν θα έπρεπε να δεχτούμε μια κατάσταση κατά την οποία εμείς οικοδομούμε σχέσεις με χώρες, αυτές που αναφέρατε εσείς, και βασιζόμαστε στον χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Δεν θα λειτουργήσει αυτό. Εάν πιστεύουμε πως θα έρθει κάποια στιγμή ξαφνικά αυτό το λαμπερό μέλλον που περιμένουμε, νομίζω ότι αυτό είναι μια αυταπάτη. Οι χώρες αυτές δεν θα αλλάξουν και τι βλέπουν γύρω τους. Κακά παραδείγματα. Τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες χώρες. Και μαθαίνουν από τη γειτονιά τους. Δηλαδή αποτελούν η μία κακό παράδειγμα για την άλλη. I would in having certain political conditionality for ratifying those. Εγώ θα έλεγα πολιτική ερασιμότητα πριν την επικύρωση αυτών των συμφωνιών. Διαφορετικά δεν θα έχουμε πια κανένα όπλο για να μπορούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να ζητήσουμε να προοδεύσει κάπως η κατάσταση. Μπορεί να συνεδριάζουμε κάθε τόσο, αλλά φοβάμαι πως οι εκθέσεις που θα λάβουμε από τους εμπειρογνώμονες που θα καλέσουμε θα είναι οι ίδιες, σε μεγάλο βαθμό. Να σας πω πως την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, οι συνάδελφοι και εγώ θα κάνουμε ένα γύρο τραπέζης για να τιμήσουμε την επέτειο της φαγής του Αντιζάν και εκεί θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε την κατάσταση στο Ουσμπεκιστάν σε βάθος για να δούμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η Human Rights Watch και οι αντιφρονούντες πώς θα επιβιώσουν όταν έχουμε τέτοια με τα σοβιετικά καθεστώτα. Συμφωνώ μαζί σας. Μπορεί κανείς αυτούς τους, ε, αυτούς τους πράκτορες θα τους βρείτε παντού. Και στο πιο απομακρυσμένο χωριό αυτών των χωρών. Πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να επιβιώσουν, πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε. Very uh, Uh, Αυτό θα ήθελα να μου πείτε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λοκπίλερ. I think if I remember right, also our AFET committee. Αν θυμάμαι καλά, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ετοιμάζουμε μία έκθεση για την Κεντρική Ασία, οπότε πολλά από τα θέματα που συζητάμε και από τις συστάσεις που έχουμε εδώ μπορούν να τοποθετηθούν σε εκείνη την έκθεση. Τρεις ερωτήσεις έχω να κάνω. Καταρχήν, Μία για το Ουσμπεκιστάν. Για την κυρία Τάγεφ. Είπατε πως όσοι ε, μιλούν για την υποχρεωτική δουλεία ε, στο χώρο της ε, συλλογής Βάμβακος αντιμετωπίζουν περιορισμούς όταν προσπαθούν να βγουν από τη χώρα. Τι συμβαίνει αυτό, υπάρχουν και άλλοι αντιφρονούντες που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Πιστεύετε πως θα ήταν χρήσιμο οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αλλά και κάποιες υπηρεσίες του ΟΗΕ στην Τασκέντε να συναντώνται δημόσια με τους ανθρώπους αυτούς για να δείξουν ότι τους στηρίζουν. Εσείς τι προτείνετε. Η, Ευρωπαϊκή, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να κάνει επιτόπια για να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών. Για το Τουρκμενιστάν Τα όσα είπατε με οδηγούν στο να πιστεύω πως τώρα θα ήταν η σωστή στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντατικοποιήσει τις επαφές που έχει με εξωματούχους από το Τουρκμενιστάν γιατί δεν θέλουν να έχουν αυτές τις μονοπωλιακές σχέσεις με την Κασπρόμ. δεν γίνεται διάλογος για ανθρώπινα δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Γίνεται με τη χώρα αυτή. Οκ, ίσως δεν σας κατάλαβα. Η ερώτηση λοιπόν πηγαίνει προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Στην απάντησή σας δεν συζητήσατε το θέμα αυτό, δηλαδή... Είπατε, χρειαζόμαστε μια συμφωνία εταιρική σχέση. Αλλιώ θα μείνουμε εκτό. Αλλά δεν θεωρείτε κι εσεί πω αυτή τη στιγμή έφτασε η ώρα να απαιτήσουμε ε, βελτιώσεις, για παράδειγμα, ε, για τις ε, υποχρεωτικές καταναγκαστικές εξαφανίσεις, όπου ξέρει η κυβέρνηση που βρίσκονται οι άνθρωποι, δεν είναι πραγματικά αγνοούμενοι στη ζούγκλα και να απαιτήσουμε πως θα έχουμε κάποια πρόεδρο. Και τέλος, για την εξωτερική δράση επίσης, υπήρξε εξωτερική δράση για το Καζαχστάν, είπατε πως εκτός από το Κυργιστάν δεν βλέπετε να υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Αλλά σε μια δήλωση πριν από μερικές μέρες, τον Απρίλιο για το Καζαχστάν, είπατε, εν πάση πτώση ο εκπρόσωπό σα στην υπηρεσία εξωτερική δράση, είπατε πω αυτή τη στιγμή είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη στήριξη έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τι περαιτέρω μεταρρυθμίσει που θα ενισχύσουν τη δημοκρατία στο Καζακστάν. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα βήματα για να ενισχύσουν τη δημοκρατία περιπτώσει, μην τη χαρακτηρίζετε δημοκρατία, δεν νομίζω πως ε, σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντα ε, του ομιλητέ μα που είναι σήμερα παρόντε εδώ και για τι εισηγήσει του που ήταν εξαιρετικά πολύτιμε και σημαντικέ. Βεβαίω υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τους ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αλλά εγώ θα ήθελα να δούμε καλύτερα τι κάνουμε εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Μπορώ να κατανοήσω σε κάποιο βαθμό την ανάγκη για διπλωμα, χρήση διπλωματικής γλώσσας στις σχέσεις με άλλες χώρες, όμως εμείς το Κοινοβούλιο, ως μέλη αυτού του Κοινοβουλίου, πιστεύω ότι πρέπει ότι μάλλον χαίρουμε πολύ μεγαλύτερης ελευθερίας έκφρασης όταν συζητάμε με τις αρχές άλλων χωρών και από όσο γνωρίζω από όλες τις δημοσκοπήσεις οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν συμπαθούν καθόλου τα αυταρχικά καθεστώτα ή τις ε, δικτατορίες. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, ε, προτάσεις ως συνέχεια αυτής της ακρόασης θα έλεγα γιατί διαφορετικά αυτό η ακρόαση θα μείνει εδώ με αυτά μαζί μας, με αυτά που μάθαμε αλλά ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Καταρχήν Μιλάμε βέβαια και λέμε ότι πρόκειται για την Κεντρική Ασία, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε χώρα είναι ε, μια χώρα ξεχωριστή με τις δικές της αποχρώσεις ε, ε, περιθώριο ευκαιρίας για να αρχίσει διάλογος με τις αρχές και γι' αυτό η πρότασή μου ως συνέχιση αυτής της εκρόσης ήταν να στείλουμε επιστολές σε κάθε μια από τις κυβερνήσεις κάθε χώρας στην Κεντρική Ασία εξηγώντας ότι έγινε αυτή αυτή ακρόαση. Δεν θέλω δηλαδή να βασιστώ μόνο στα όσα τα μέλη των διαφόρων ε, πρεσβειών θα θελήσουν να τους διαβιβάσουν. Εμείς να μπούμε σε διάλογο με τις κυβερνήσεις, να πούμε ότι κάναμε αυτήν την ακρόαση, να πούμε ότι ανησυχούμε για διάφορα ε, ζητήματα και βεβαίως ε, ότι υπάρχουν προβλήματα για όλες τις χώρες αυτές. Αλλά να πούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι η κύρια μας προτεραιότητα είναι να σώσουμε ζωές σε αυτή την, εδώ την Επιτροπή. Ίσως λοιπόν ε, ονοματίζοντας τους ανθρώπους που είναι στις φυλακές να μπορέσουμε να, κάνουμε, να σημάνουμε τη διαφορά ευγενικά, πολιτισμένα, αλλά πολύ ε, ε, σταθερά και επίμονα ταυτόχρονα. Αυτή είναι η πρότασή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλή η πρότασή σας. ξέρω αν η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θέλει να πάρει το λόγο για να απαντήσει κάτι στις ερωτήσεις που έκανε η κυρία Λοκμπίλερ. Μήπως θέλετε. First of all, maybe starting with the last comments, I... Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο σχόλιο. Στηρίζω απολύτως αυτή την ιδέα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει να, να αναλάβει πιο έντονη δράση σε σχέση με το θέμα της ε, Κεντρικής Ασίας και να στηρίξει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και στις χώρες αυτές. Είναι δεδομένο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πολύ παρούσα στην Κεντρική Ασία, δηλαδή με την εξαίρεση του Καζαχστάν έχουμε ελάχιστες πρεσβείες των κρατών μελών και οι πρεσβείες αυτές είναι μάλλον μικρές συνήθως. Εάν θέλουμε λοιπόν να είναι πιο έντονη η παρουσία μας, θα πρέπει να είμαστε και σωματικά παρόντες. για το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν, Να ξεκινήσω με το Καζακστάν, λέγοντάς σας πως είχαμε κάποια θετικά στοιχεία στις πρόσφατες εκλογές που στη χώρα, η διοργάνωση των εκλογών ήταν αρκετά αποτελεσματική. Βέβαια ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι να θεωρηθούν ελεύθερες και δίκαιες αυτές οι εκλογές και εμείς ασκήσαμε πολύ κριτική για το θέμα αυτό. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μόνιμο συμβούλιο του ΑΣΕ επαναλαμβάνονταν εξαιρετικά επικριτική και μιλήσαμε για τους παρατηρητές του ΑΣΕ που αντιμετώπισαν πολλές διαδικαστικές δυσκολίες και παρατυπίες. Όμως είδαμε πως υπάρχουν βήματα πρόοδου και θα θέλαμε να στηρίξουμε το Καζακστάν στο να προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι δύσκολη η περιοχή αυτή και γεωπολιτικά. Έχουμε την Ρωσία, την Κίνα. Δεν είναι εύκολη περιοχή για να πλοηγηθεί κανείς με ασφάλεια. Και από τις τρέχουσες οικονομικές ε, συνθήκες όπου αρκετές χώρες Κεντρικής Ασίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες, η πρώτη τους αντίδραση, η αντανακλαστική, μοιάζει να είναι να περιορίσουν τις αρνητικές απόψεις, επειδή ακριβώς φοβούνται ταραχές και εσωτερική αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να παραμένουμε στο παιχνίδι και θεωρούμε πως έτσι δεν παραδίδουμε αμαχητή την ευθύνη μας ε, στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι. Μιλάμε για αυτά και θα συνεχίσουμε να τα θίγουμε και για το Τουρκμενιστάν εκεί δεν υπάρχει πολιτικός διάλογος. Δεν γίνεται καμία συνάντηση σε υπουργικό επίπεδο, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε επίπεδο υψηλών ανώτατων αξιομετούχων. Τώρα, εσείς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους τουρκμένους βουλευτές, αλλά ίσως εκεί θα έπρεπε να βρείτε το τρόπο να περάσετε το μήνυμά σας. Εάν δεν έχουμε τέτοιες διαδρομές συζήτησης, το να ελπίζει κανείς στο ότι απλώς θα αλλάξει κατάσταση είναι δύσκολο. Είναι σημαντικό να μιλάμε Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικέ εξελίξει. Σε πολλέ περιπτώσει δεν είναι, αλλά η εναλλακτική λύση είναι να αποσυρθούμε από το διάλογο αυτό και δεν θεωρούμε πω με τον τρόπο αυτό θα καταφέρνουμε οτιδήποτε. Για πολύ λίγο χρόνο θα δώσω στους προσκεκλημένους μας το λόγο και θα πάμε από την άλλη μεριά. Ξεκινάτε εσείς στην άκρη για δύο λεπτά. <clears throat> Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ε, πρέπει να είμαι τελείως τηλεγραφικός παρά το ότι όλα αυτά αξίζουν βεβαίως ε, συζήτηση. Ε, πρώτα απ' όλα θεωρώ πως είναι λάθος το δίλημα. Το θέμα δεν είναι επιλογή μεταξύ της μη επαφής ή της επαφής ανεφόρων. Είναι ψευτοδίλημα. Εμείς ε, θεωρούμε πως η αιρεσιμότητα αυτή δεν λειτουργήσε γιατί δεν εφαρμόστηκε σωστά και δεν ήταν σωστή η όρη. Το συζητήσαμε και υπάρχουν ε, πολύ περισσότερα στοιχεία τώρα που δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε λεπτομερώς ε, όσον αφορά την συμπεριφορά συγκεκριμένων διπλωματικών εκπροσώπων στο Τουρκμενιστάν που επιδεικνύουν τρομερό ενδιαφέρον ε, και δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν και τώρα έχουμε αυτό το μοχλοποίηση. Δεύτερον, εμείς δεν ζητάμε απομόνωση. Αντιθέτως, ζητάμε μία εμπλοκή η οποία θα είναι ενεργός και επικριτική, χρησιμοποιώντας του, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για πίεση. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτά μπορεί να είναι περιοριστικά μέτρα, όπως στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, αλλά αυτό είναι άλλο. Δεύτερον, υπήρξε ένα συγκεκριμένο ερώτημα για τον ρόλο της Επιτροπής Ασφαλείας ε, του Τουρκμενιστάν το εάν είναι ένα μέσο παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, οπωσδήποτε, όπως σε οποιοδήποτε αυταρχικό καθεστώς ή χώρα με δικτατορία, η υπηρεσία ασφαλείας είναι το βασικό κομμάτι καταστολής. Όλο το σύστημα είναι κατασταλτικό και η υπηρεσία ασφαλείας είναι σημαντικό κομμάτι. Πώς επιζούν οι ακτιβιστές πώς μπορεί να τους στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό ερώτημα. Πολλοί από αυτούς, όπως ξέρετε, αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα. Ε, αρκετοί βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Δεν μπορούν να είναι πλέον στη χώρα τους και να δουλέψουν ανοιχτά και χωρίς φόβο διώξεων. Άλλοι έχουν αφήσει πίσω συγγενείς. Και είναι ευάλωτοι και εκτός της χώρας όταν φεύγουν και είναι σε αυτοεξορία ε, και εκεί τους στοχεύουν οι μυστικές υπηρεσίες. Αυτό έγινε πάλι και με κάποιους που είναι σε αυτή την αίθουσα. Είναι μεγάλο λοιπόν το θέμα. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τακτικούς διαλόγους ε, και επαφή σε ένα περιβάλλον ασφαλές. Τώρα δεν υπάρχει μία συνταγή για αυτά τα θέματα, αλλά από μπορώ να πω για το Τουρκμενιστάν δεν υπάρχει επαφή μεταξύ του Γραφείου Συνδέσμου της Ένωσης και ανεξαρτήτων ε, ακτιβιστών. Μεμονωμένων ατόμων, ναι, αλλά ακτιβιστών τώρα δεν ξέρω. Τώρα, Τώρα για τη σημασία της ε, παρουσίας μας εκεί επί τόπου. Ναι, πράγματι έχει σημασία η επαφή, πράγματι, και δεν λέμε αναβολή επαόριστον. Αλλά να έχουμε τώρα άμεση επαφή, να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα και να πάμε σε μία μη δομημένη, αν θέλετε, εμπλοκή με σαφή προοπτική της ε, κύρωσης σε, μισό, σε έξι μήνες, ένα χρόνο, αν υπάρχει αυτή η πρόοδος. Υπάρχουν τρόποι να γίνουν αυτά. Και ακόμα και το να ανοίξουμε μια αντιπροσωπεία είναι δυνατόν ακόμα και απουσία συμφωνίας ε, σύνδεσης. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Θα ήθελα κι εγώ εκ μέρου πολλών συναδέλφων που δεν μπορούσαν να είναι εδώ σήμερα καταρχήν να εκφράσω τις τεράστιε τις ευχαριστίες μας γιατί και την προηγούμενη φορά που μας καλέσατε ε, μιλήσαμε εδώ για το θέμα της παιδικής εργασίας καταναγκαστικής στο Ουσβεκιστάν να σας πω πως το θέμα αυτό ε, ξέρετε πως δεν έχει εξαφανιστεί αυτό το φαινόμενο εκτός ε, πρωτεύουσα εξακολουθεί να υπάρχει όχι βέβαια τόσο μαζικά όσο στο παρελθόν αλλά προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και έχουμε το εξής πρόβλημα η κυβέρνηση του Ουσμπεκστάν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσφέρει ε, εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά της χώρας και είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. Ελπίζω πως το νέο στρατηγικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουσμπεκιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ε, μας επιτρέψει να δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και να ληφθούν όντως υπόψη. Θα ήθελα επίσης να σας πω πόσο χάρηκα που εσείς είπατε πως θα απευθυνθείτε ε, με επιστολές στην ε, κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το να στείλετε εσείς ε, επιστολές με συγκεκριμένους ε, κρατουμένους πιστεύω πως θα επηρεάσει την κατάσταση και θα δώσει κάποιο αποτέλεσμα. Για το Μουράτ να σας πω πως 21 χρόνια κρατείτε και την τρίτη καταδίκη ε, για, που καταδικάστηκε για τέσσερα χρόνια φυλάκιση είναι γιατί δεν καθάρισε καλά τα καρότα στη φυλακή. Το καταλαβαίνετε αυτό είχε απαχθεί από το Καζακστάν ε, κρατήθηκε στις δικές μας φιλικές και να σας πω πως το Δεκέμβριο στο Ουσμπεκιστάν έγινε και μια δίκη Ενα, καταδικάστηκαν οκτώ ε, πολίτες που μετά ε, απελάθηκαν στον, στην Ορβηγία και ένας από αυτούς η γλώσσα του την είχαν ισχύσει στα δύο. Δυστυχώς ούτε η Νορβηγία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε οποιαδήποτε δήλωση, ε, ούτε αναφέρθηκε για κανείς σε τεκμήριο αθωότητας. Είμαστε στον 21ο αιώνα ε, και καταδικάζονται άνθρωποι σε βασανιστήρια σαν να βρισκόμαστε στη δεκαετία του 30. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν δυνατότητα ε, έφεσης στις περιπτώσεις αυτές. Άρα λοιπόν η φωνή των δημοκρατών από την Ευρώπη θα είναι για μας μια πολύ σημαντική στήριξη. Να σας υπενθυμίσω πως η Λετωνία κάλεσε τον κύριο Καρίμοφ σε κάποιες εκδηλώσεις και αυτό ανισχύει πάρα πολύ τον ουσβεκικό λαό γιατί αυτός διάταξε τους πυροβολισμούς που σκότωσαν κόσμο στο Ιντιζάν και καταλαβαίνετε πως το να τον προσκαλείτε είναι ανισχυτικό. Θα ήθελα να κοιτάξετε και το εξή. Στο Ουσβεκιστάν, εδώ και ένα χρόνο παρόνομα, έχουμε παραπάνω από 100 πρόσφυγες από την κοιλάδα του ΟΣ. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στο Ουσβεκιστάν χωρίς να έχουν χαρτιά, το Δεκέμβριο χάσανε, τους έκλεψαν τα διαβατήριά τους, τους πήραν μάλλον τα διαβατήρια και είναι τα θύματα μιας εθνοτικής σύγκρουσης. Δεν έχουν καταγραφεί πουθενά ε, έφυγαν ε, από τον Κυργιστάν, βρήκαν καταφύγιο στο Ουσμπεκιστάν και με μια μυστική συμφωνία για την ανταλλαγή προσφύγων το Ουσμπεκιστάν με μυστικό τρόπο έχει, έχει υποσχεθεί στη χώρα που απειλεί τη ζωή τους να τους στείλει πίσω σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν μια δίκαιη δίκη και για τους αντιφρονούντες από το Καραπα... Καλβαστάν ε, υποσχέθηκε πως θα τύχουν αντίστοιχες μεταχείρισεις επίσης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως αυτή τη στιγμή έχουμε μυστικές επισκέψεις από αξιωματούχους του Ουσμπεκιστάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κεντρική Ασία. Πιστεύω πως αν τους απαγορευτούν αυτές οι επισκέψεις θα έχετε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία παρά αν συνεχίσετε με αυτές τις μυστικές επαφές που έχετε. Υπάρχουν ακτιβιστές οι οποίοι κινδυνεύουν. Ε, κινδυνεύει η ζωή τους, ε, κινδυνεύει η σωματική τους ακαιρεότητα. Θα ήθελα λοιπόν να τους βοηθήσουμε και σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Έχω uh, πολύ σύντομες παρατηρήσεις η μία φορά τις εκλογές. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, ε, είπατε, στις εκλογές. Μα δεν ήταν εκλογές αυτές. Αλλιώς ε, να λέμε ότι και οι εκλογές στην Έσουσουδού ήταν καλά οργανωμένες από την τεχνική σκοπιά. Μα δεν ήταν εκλογές αυτές. Πράγματι, ξαναβγήκε ο πρόεδρος Ναζαρμπάγεφ, αλλά εκλογές σημαίνει πλουραλισμό. Να υπάρχει χώρος για την αντιπολίτευση και να επιτρέπεται στους ε, πολιτικούς να αναπτύξουν λόγο, να έχουν πρόσβαση στα πανεθνικά μήμια. Αυτό δεν θα γίνει, ανεξαρτήτως του τι κάνει η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Ειδικά όταν έχουμε γεγονότα ότι πηγαίνει κόσμος ε, με τα πούλμαν στα εκλογικά κέντρα. Αν δεν υπάρχει δηλαδή μια προεκλογική περίοδος πλουραλιστική δεν μπορούμε να, έχουμε, να μιλάμε για δημοκρατία. Μετά, το πώς επιζούμε. Αυτό διαφέρει ένα χώρο. Στο Τουρκμενιστάν, όπως είπε ο Γιούρι, δεν επιζούν, εξαφανίζονται οι άνθρωποι, είτε στη φυλακή είτε στην εξορία. Το ίδιο σε ένα βαθμό και για το Ουσβέκισταν και το Τατζικιστάν. Κα, Καζακστάν και Κυργιζία. Λιγότερο επικίνδυνες χώρες, μας παρακολουθούσαν ε, τα τηλέφωνα και τα λοιπά, αλλά και πάλι είναι μια ήπια τρομοκρατία. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο είπε ο Γιούρι. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτύχει θετικά αποτελέσματα, όπως σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως το Ουσπεκιστάν και το Τουρκμανιστάν περιμένουμε... Τι, ναι, τι περιμένουμε. Τουλάχιστον πρόσοχη, μια ηθική στήριξη, τη στήριξη του διαλόγου με την ε, κυβέρνηση που βελτιώνεται όπως είπαμε στο Καζακστάν κάπως και να παρακολουθούμε συγκεκριμένα την κάθε περίπτωση. Γι' αυτό ε, και η περίπτωση των τριών πολιτικών κρατουμένων. Τέλος για αυτούς που είναι σε ε, εξορία. Εδώ πέρα δηλαδή πραγματικά γίνεται κατάχρηση της Interpol. Πρέπει να το δει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς χρησιμοποιούν οι χώρες αυτές την Interpol για να διώκουν ε, τους αντιπάλους τους και στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο για Καζάκους, αλλά και για Ουσμπέκους και άλλους. Και στην Ευρώπη ακόμα. Και είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δηλαδή, τι θα κάνει η Interpol να είναι κάπως πιο προσεκτική ειδικά να χρησιμοποιήσει τα κριτήρια της ύπα αρμοσίας για τους πρόσφυγες, γιατί πολλοί από αυτούς αναζητούν άσυλο στην Ευρώπη. Νομίζω πως ε, θα, έχουμε θετικά, θα μπορούσαμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποια σύντομα σχόλια για τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρούν πως είναι σημαντικός ε, για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων, αλλά εμείς ε, θα θέλαμε να ενισχυθεί ως ένα εργαλείο που θα έχει θετικά αποτελέσματα. Με το να έχουμε σαφείς στόχους ε, γίνεται σαφής και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το να ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο του διαλόγου υπάρχει κάποιο, κάποιο, υπάρχουν κάποια επίσημα πρακτικά. Βεβαίως αν δίνεται συνέχεια και ειδικά στο υψηλότερο επίπεδο υπάρχει δυνατότητα να γίνει γνωστό και το περιεχόμενο του διαλόγου. Όταν μιλάμε τώρα για ενισχυμένες σχέσεις με Τουρκμενιστάν και Καζακστάν, μιλάμε για μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για να ζητήσουμε συγκεκριμένες και μετρήσιμες μεταρρυθμίσεις ε, στο Τουρκμενιστάν. Αυτά έγιναν από το Κοινοβούλιο το 2008 και επαναβεβαιώθηκαν το 2010 απελευθέρωση δηλαδή πολιτικών κρατουμένων, άρση απαγόρευσης ε, ταξιδιού στο εξωτερικό, να επιτραπεί ε, είσοδος στη χώρα παρατηρητών του ΟΗΕ. Πρέπει να γίνουν αυτά πριν ε, καταλήξουμε επιτυχώς στις διαπραγματεύσεις Παραμία στο Καζακστάν. Και εδώ πέρα η υπηρεσία εξωτερική δράση είπε πω θα ήθελε να στηρίξει το Καζακστάν. Μπορεί να το κάνει αυτό με το να έχει σαφεί προσδοκίε για μεταρρύθμιση. και βεβαίως έτσι θα έχουν νόημα και αυτά τα οποία ε, είπε η Κάθριν Άστον και τα ψηφίσμα του Κοινοβουλίου το 2012 και 2013. Για το Ουσμπεκιστάν, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, πρέπει να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, των Υπουργών δηλαδή, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλιώς θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες συνέπειε. Και τέλο το τι γίνεται για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ θα επανέλθω στις συστάσεις που κάναμε για το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να οθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση. Και για το ότι δεν υπάρχει χώρος στην κοινωνία των πολιτών να πιέσει τις κυβερνήσεις να επιτρέψουν την ειρηνική αντιπολίτευση και να δουν τον νόμο περί ξένων πρακτόρων στην Κυργυζία για τη στήριξη των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά ε, αυτών που βρέθηκαν στη φυλακή. Και εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις σε ολόκληρη την ε, Κεντρική Ασία και το να τους κατανομάζουμε είναι κάτι σημαντικό. Και τέλος, η πρόσβαση για τους μηχανισμούς του ΟΗΕ ειδικά στο Ουσβεκιστάν και το Τουρκμενιστάν όπου υπάρχουν ε, γύρω στους 12 μηχανισμούς που δεν έχουν μπορέσει να έχουν πρόσβαση στη χώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ανταλλαγή απόψε και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ναι, αναμένετε το αποτέλεσμα. Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια συνέχεια και υποθέτω έχοντας ακούσει και τους τέσσερις σας ε, και την κατάσταση στις χώρες όσοι οι παραβιάσεις αυτές είναι τόσο σοβαρές που οπωσδήποτε θα μας απασχολήσουν ξανά είχαμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Τουρκμενιστάν και οπωσδήποτε και οι επισκέψεις της ε, ΑΦΕΤ ε, θα αποτελέσουν άλλη μια ευκαιρία σας ευχαριστώ λοιπόν και καλή δύναμη για την συνέχεια και συνεχίστε να παλεύετε κατά του αυταρχισμού. Okay, colleagues, could we start, please? μπορούμε να ξεκινήσουμε. Με το επόμενο θέμα και παρακαλώ οι συζητήσεις εκτός της ε, αίθουσας.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 Παρακαλώ οι συζητήσει εκτός της αιθούση. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο. Μια προσέγγιση της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία, το ευρωπαϊκό κληροδότημα για τη δημοκρατία. Έχουμε μια έκθεση εδώ του εισηγητή μας, του κυρίου Σιπ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη δουλειά που κάνατε στις ε, τροπολογίες. Έχετε λάβει 104 ε, τροπολογίες, ε, οπότε ήταν δύσκολη η δουλειά σας. Νομίζω λοιπόν πως τώρα μπορούμε να συζητήσουμε την έκθεση. Επίσης η ψηφοφορία είναι στις 26 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος. Και στις 13 Μαΐου Υπάρχει άλλη μια συνεδρίαση των σκιωδών στις Βρυξέλλες. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βλέπω τους κυρίους Dennis Μάκερ. ο κύριος Λίτς αντικαθιστά τον κύριο Μάρτιν από σοσιαλδημοκράτες και ίσως έρθουν και άλλοι. Κύριε Ζιμπ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήδη είπατε αρκετά από αυτά τα οποία έπρεπε να υποθούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που τονίζετε το ότι έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες, πόσες τροπολογίες έχουν υποβληθεί και ποιος είναι ο σκιώδης ε, εισηγητής. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, και να εξηγήσω πως κάποιες από αυτές τις τροπολογίες είναι κοινέ ε, τροπολογίες που υποβάλαμε μαζί με τους συναδέλφους. Υπέβαλα λοιπόν κάποιες ε, τροπολογίες για τους εξή λόγους. Ενώ προετοίμαζα το σχέδιο έκθεσης λόγω των περιορισμών στον αριθμό λέξεων δεν μπόρεσα να βάλω κάποια πράγματα και άρα τα παρέλειψα. Αλλά επειδή είναι τόσο σημαντικά, αποφάσισα ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Οπότε υπέβαλα και εγώ κάποιες τροπολογίες γιατί προέκυψαν και από την συζήτηση που, που ξεκίνησε αφού υπέβαλα το σχέδιο συζήτηση με οργανώσεις, φορείς που εμπλέκονται άμεσα στην χρήση του ευρωπαϊκού αυτού κληροδοτήματος για την δημοκρατία αλλά και συζήτηση με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με την Κομισιόν αλλά και με τους συναδέλφους εδώ πέρα από διάφορες ε, πολιτικές ομάδες που διάβασαν την έκθεση και είπαν πως έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους με τους οποίους υπέβαλα κάποιες κοινέ τροπολογίες, ειδικά τον κύριο Μισελ και την Αλεξάνδρ Λαφίν Στότ, τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπιουτικόφερ, τον σκιώδη τους συναδέλφους από το ΕΛΚ, ειδικά τον Έλμαρ Μπρόκ, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, Εξωτερικών και τον Κρίστιαν Πρέντα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Ντέιβιντ Μάρτιν για την θετική του συνεισφορά στο κείμενο, ειδικά την τροπολογία υπαριθμών 99 ζητάει από το κληροδότημα να αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους για να στηρίξει την δημοκρατία. Οπουδήποτε λοιπόν υπάρχουν περιορισμοί στην δημοκρατία. Οπότε τονίζει τις βελτιώσεις ε, που μπορούν να γίνουν και τον ρόλο που πρέπει να παίξουν τα νέα μέσα είναι μια βελτίωση νομίζω που μπορεί να γίνει. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμέσμα επειδή στηρίζει πλήρως το σχέδιο το οποίο πρότεινα. Υπάρχουν και τροπολογίες που πρότεινε το ECR, ο κύριος Τζαμπάσκι. Ειδικότερα θα ήθελα να τονίσω μια τροπολογία η οποία επικεντρώνεται στην ε, εμπειρία που έχουμε στις χώρες εκείνες που είχαμε την δημοκρατική μετάβαση. Και η εμπειρία έχει δείξει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η μετάβαση για να θέσουμε στόχους και πάλι ο κύριος ε, Ιγνάσιο Κοράου ε, σκιοδησηγητή συζητάει από τα κράτη-μέλη να στηρίξουν ε, την μεταρρύθμιση αυτή. Γνωρίζουμε πως οι στόχοι μας εξαρτώνται από τις οικονομικές συνεισφορές ε, πλην βεβαίως των διοικητικών εξόδων. Οπότε ε, οι δωρεές καλύπτουν απευθείας τις δραστηριότητες του κληροδοτήματος. Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Κάποιες από αυτές τις τροπολογίες μιλάνε για πολιτική αντιπροσωπευτικότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι βεβαίως προνόμιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κληροδότημα δεν έχει την δυνατότητα να επηρεάσει τις αποφάσεις του ΔΣ. Πρόκειται λοιπόν για έναν νεότατο οργανισμό και καθώς προχωράει το έργο κερδίζει και σε εμπειρία το Ίδρυμα και καθώς προετοίμαζα το σχέδιο έκθεσης ε, υποστήριζε το κληροδότημα γύρω στα 127 έργα με, ε, ένα, ενώ έχουμε φτάσει πλέον ε, στα 8 εκατομμύρια ευρώ και 143 έργα. Αυτό δείχνει πως ο χρόνος δουλεύει υπέρ ημών, όπως και η πολιτική μας συντολή, η οποία επεκτείνεται. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα συμπεριλάβω, δεν μπορώ να συμπεριλάβω και να στηρίξω όλες τις τροπολογίες. Αλλά αυτή η εξαίρεση ισχύει για λίγες από τις 104 ε, τροπολογίες. Να δώσω ένα παράδειγμα μίας τροπολογίας όμως, η οποία προτείνει να διαγραφεί μια φράση. Δηλαδή, η φράση που μιλάει για την χρηματοδότηση γέφυρα, μια μεταβατική χρηματοδότηση. Μα αυτό ακριβώς είναι ένα κομμάτι προστιθέμενης αξίας του κληροδοτήματος ε, γιατί ακριβώς καλύπτει τη χρηματοδότηση μεταξύ των κενών. Επειδή δηλαδή η χρηματοδότηση προέρχεται από άλλους οργανισμούς και άλλα πράγματα περιγράφονται εδώ. Το σχέδιο έκθεσης μιλάει και για άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς και λέει πως ε, αρκετοί από αυτούς στρέφονται στο κληροδότημα γιατί έχει τη δυνατότητα να τους δώσει αυτή τη μεταβατική χρηματοδότηση. Λοιπόν, προτείνω πρώτη ανάγνωση 13 Μαρτίου, Τετάρτη και θα ήθελα να πω στους συναδέλφους τους και όδησης ηγητές πως προετοίμασα ήδη ένα πρώτο σχέδιο της ε, έκθεσης ε, και θα το στείλω για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτό και ελπίζω να συνεχίσουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε και θα επιτύχουμε έναν αποδεκτό συνδυασμό. Κάποιε περιπτώσει ίσως αρκεί μια προφορική τροπολογία για να είναι πλήρη η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Οι σκιώδε λοιπόν. Ο κύριο Θέμης Μακερνό Ευχαριστώ. Λίγα έχω να προσθέσω σε αυτά τα οποία μόλις είπε ο κύριος Ξύπ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ για την δουλειά που κάνατε. Να υποποστηρίζουμε σε μεγάλο, σε γενικές γραμμές την έκθεση. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που επικαιροποιούν τους αριθμούς. Αυτό χρειάζεται. και πράγματι θα δούμε κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις διάφορες παραγράφους ε, σε σχέση με την χρηματοδότηση συμπληρωματικούς δεσμούς με άλλους οργανισμούς ε, συνεργασία με θρησκευτικές κοινότητες εμείς οπωσδήποτε είμαστε υποστηρικτές των τροπολογιών που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στα δικαιώματα εθνικών μειονοτήτων. Έχουμε υποβάλει κάποιες ε, ε, τροπολογίες και θα τα δούμε αυτά μετά πιο λεπτομερώς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα συνταχθώ με τον κύριο Τένις Μάρκερ και θα ευχαριστήσω και τον εισηγητή όχι μόνο για την ε, έκθεση τη συγκεκριμένη αλλά για όσους προσπάθειες έχει κάνει τόσα χρόνια για να προοδεύσει αυτό το θέμα και να γίνει κομμάτι της πραγματικότητας υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός συνένεσης και στήριξης για το πληροδότημα αυτό, όπως επίσης και για το όλο περιεχόμενο της έκθεσης, οπότε με μεγάλη χαρά περιμένω τους ε, περιεκτικούς ε, συμβιβασμούς που μας είπατε πως θα λάβουμε κύριε Σρίπ. Μία μικροπαρατήρηση. Δεν έχετε αναφερθεί πολύ στη γεωγραφική, στο γεωγραφικό πεδίο. Ίσως μισή σελίδα να χρειάζεται. Οι 27 τροπολογίες ε, που έχουμε υποβάλει αποδεικνύουν πόσο ε, στηρίζουμε, ε, συγχωρείτε πόσο μας ενδιαφέρει το θέμα να πω το εξή. Εμείς καταρχήν δεν προσπαθούμε να αφαιρέσουμε σημασία από το κληροδότημα αυτό. Παρόλα αυτά κάνουμε κάποιες άλλες αναφορές σε άλλα ιδρύματα τα οποία στηρίζουν και αυτά με τη σειρά τους τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προτείνουμε λοιπόν κάποια φρασιολογία έτσι ώστε και, το, και τα άλλα ιδρύματα που είναι το σχετικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα να στηριχθεί γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανταγωνιστικά μεταξύ τους ε, όργανα. Επίσης, σε κάποια καρδιμέλη όπως το δικό μου, το κληροδότημα επιβαρύνεται με διοικητικές ε, ε, διοικητικό φόρτο ε, και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το αντικρούσουμε. Δεύτερον, οι προτάσεις μας, και θα θέλαμε να τις στηρίξουν και οι υπόλοιπες ομάδες, μιλάνε για τη μελλοντική δράση του κληροδοτήματος. Δηλαδή περιθωριοποιημένες μειονότητες, ε, σε περιοχές με παγωμένες συγκρούσεις, για τις εθνικές μειονότητες, τα συνδικάτα, τους αναδυόμενους νέους ηγέτες και τις νεοεκλεγόμενες γυναίκες ή εκπροσώπους μειονοτήτων. Αυτά θα μπορούσαν να προσθέσουν στο πεδίο. Επόμενη παρατήρηση. Για την παράγραφο 4 μου δημιουργεί κάποιες ανησυχίες αυτού το επισημοποιημένο, επισημοποιημένη διέρεση στη συμμετοχή μεταξύ Βορράς και Νότου. Δεν νομίζω πως τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται μόνο για την πολιτική γειτονία προς την Ανατολή ή προς, την, προς τον Νότο, ε, ανεξάρτητα με τη γεωγραφική του θέση. Και στην τροπολογία 53 προσπαθούμε αυτή την ε, φράση κάπως να την χρωματίσουμε. Και τέλος, κύριε Τζαμπάστη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. είτε τώρα είτε στο μέλλον, θα ήθελα να λάβω μια απάντηση στο εξή. Η τροπολογία 69 τι σημαίνει, γιατί μιλάμε για κατηγορίες που απευθύνονται προς προς το ε, ίδρυμα αυτό για το πληροδότημα, ε, οι οποίες δεν έχουν ε, τεκμηριωθεί. Και λέει, για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων για χρηματοδότηση από το κληροδότημα έτσι ώστε να αποφευθεί η απευθείας ή η εμεση χρηματοδότηση τρομακρατικών ομάδων ή ατόμων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ε, τη δημοκρατική διαδικασία και εκδημοκρατισμό ε, στις ε, χώρες της πολιτικής γειτονίας για τον Νότο. Μα αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί. Δεν τεκμηριώνεται πουθενά αυτή η καταγγελία. Δεν βλέπω να είναι εδώ ο συνάδελφος στον οποίο αναφερθήκατε. Νομίζω λείπει και δεν βλέπω κανέναν άλλον από τους κοιόδες. Κύριε Σρίπ, μήπως η κυρία που εκπροσωπεί την υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα μπορούσε να κάνει καμιά σχόλια και εσείς μια σύνοψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για σχόλια από τη, από τη Διεύθυνση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο συνάδελφός μου δεν είχε την ευκαιρία να σχολιάσει την περισμένη φορά. Σύντομα να σας πω ότι καλωσορίζουμε την έκθεση, συμφωνούμε με τα συμπεράσματά της και συμφωνούμε και με τις σημαντικές αλλαγές στις δυνατότητες μας να ενεργήσουμε για τον εκδημοκρατισμό μέσω της δημιουργίας ε, του Ευρωπαϊκού Κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία. Είμαστε, ε, πιστεύουμε ότι αυτό που ε, θα πράξει μπορεί να συμπληρώσει το, τα κενά, θα μπορέσει να στηρίξει τους πολιτικούς ακτιβιστές σε μεταβατικές περιόδους. Υπάρχει η παράγραφος 31, η οποία μας απευθύνεται και είναι μια επιχειρησιακή παράγραφο, απευθύνεται σε εμά το ρόλο μας ε, και στην απόπειρά μας να αυξήσουμε τη συνέπεια ανάμεσα στη ε, στάση των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Αυτό ήδη το κάνουμε. Εμεί στις υπηρεσίες της Κομισιόν και της Εξωτερικής ε, Υπηρεσίας ε, προσπαθούμε να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση σε κάθε χώρα και να υπάρχει καλύτερη ροή στις δραστηριότητές μας. Ευχαριστώ. Κύριε Ξύμπ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Να αρχίσω από το τελευταία παρατήρηση ίσως. Νομίζω πως ε, αυτό είναι ένα κίνητρο για να συνεχίσουμε με την προσπάθεια που ξεκινήσαμε να εθαρρύνουμε άλλους να βελτιώσουν την εξωτερική μας εκπροσώπηση στις τρίτες χώρες, να ενθαρρύνουμε τον εκδημοκρατισμό στις χώρες αυτές. Επίσης, ε, Πρόκειται για μια ενθάρρυνση λοιπόν ώστε οι δικαιούχοι να μάθουν ότι μπορούν να υποστηριχθούν από κάποιον. Συμφωνώ με το όσο είπε ο κ. Μπουτικόφερ μάλιστα, ότι δηλαδή θα πρέπει να τονίσουμε αυτή την ε, τροπολογία Η διατύπωση αυτή είναι κάπως ε, προκλητική. Αρκετά προκλητική. Φαίνεται να ξεχνάμε τους δυνητικούς ε, δικαιούχους που θέλουμε να στηρίξουμε και που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό το ε, κληροδότημα. Αυτή η τροπολογία είναι μία από, αυτές, από αυτά τα παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκα. Κάποιες από τις λίγες τροπολογίες που δεν υποστηρίζω εγώ. Τώρα όσον αυτά τα σχόλια που εν γέννη αφορούν την ποιότητα των διαφόρων σωμάτων ή θεσμών που λειτουργούν, την, την έλλειψη ανταγωνισμού, δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στην ΕΕΔ και άλλους ε, θεσμούς. Είναι σημαντικό και είναι κάτι το οποίο έχω τονίσει επανειλημμένως και νομίζω το κάλυψα στην εισαγωγή που έκανα. Πρέπει να φτιάξουμε σχέσεις και να δίνουμε έτσι κάποια μεταβατική χρηματοδότηση ώστε να στηρίξουμε τη δραστηριότητα εκείνων των σωμάτων που θέλουν ε, την, και χρειάζονται την υποστήριξη. Συχνά έχουμε συζητήσει στην υποεπιτροπή μας ότι Η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ε, υπάρχει, αλλά ε, ε, φέρει πολλές δεσμεύσεις και γι' αυτό και καθυστερεί. Πολύ συχνά οι επιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμες. Μπορεί όμως αυτές να μην υπάρξουν λόγω της έλλειψης κάποιων μεταβατικών δανείων, δανείων για αυτές τις μεταβατικές περιόδους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τόσο είπατε. Ελπίζω πως ε, θα μπορέσω να εντάξω τις τροπολογίες των σκιωδών με ικανοποιητικό τρόπο. Σας ευχαριστώ κύριε Ξύμπη και κατάλαβα από τη σημερινή συζήτηση. Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε, αλλά... Δεν έχουμε πρόβλημα γιατί η ψηφοφορία στις 26 Μαΐου θα γίνει, έτσι. Θα τα καταφέρετε. Ωραία, είστε έτοιμος. Πολύ ωραία. Οπότε τότε νομίζω ότι εδώ τελειώνει η δημόσια μας συζήτηση. Και τώρα θα συνεχίσουμε με συνεδρίαση κυκλισμένων των θυρών, ώστε να δούμε διάφορα κατεπήγοντα θέματα. Όλοι όσοι λοιπόν δεν ε, ε, συμμετέχουν στην συνεδρίαση κυκλισμένων των θυρών, παρακαλώ να ε, εγκαταλείψουν.